Καλημέρα, άρχεται η συνεδρίαση. Eh, e Καλωσορίζω το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το πρώτο θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι οι δηλώσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Υπουργό του Περάινεν εξ ονόματος του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο κύριε του Περάινεν. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, για μια ακόμη φορά θα συζητήσουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μια δύσκολη στιγμή και πολλοί είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που υποφέρουν από την αβεβαιότητα. Τον Ιούλιο ο νέος Πρωθυπουργός ε, που δεν βοήθησε τελικά να ξεκαθαριστεί η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου όταν ε, υπάρχουν τα δύσκολα θέματα όπως τα Ιρλανδικά σύνορα το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει καταθέσει νέες προτάσεις και οι απόψεις στο Κοινοβούλιο στο Λονδίνο ε, είναι πάντα συγκεχημένες και δεν υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά η Βρετανική κυβέρνηση επιμένει στις κόκκινες γραμμές. Η 31η Οκτωβρίου λοιπόν πλησιάζει και δυστυχώς υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Αυτή η σκοτεινή κατάσταση δεν θα πρέπει να μας απομακρύνει από τις βεσικές μας προτεραιότητες, κυρίως από ε, την τακτική αποχώρηση της συγκεκριμένης χώρας. Γι' αυτό πιέζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να μας κάνει συγκεκριμένες ορθολογικές και ακριβείς προτάσεις ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και το θέμα της απουσίας πιθανώς σκληρών σε εισαγωγικά συνόρων, σταθερών συνόρων ε, στην Ιρλανδία. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Westminster και η έκκληση για περαιτέρω παράταση ε, κάνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Πρέπει να το παραδεχθούμε ότι αυτή τη στιγμή μία μη συμφωνία για τις 31 Οκτωβρίου είναι το πιο πιθανό γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο επαναλαμβάνει συνεχώς ότι είναι διατεθειμένο να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι οι προετοιμασίες θα πρέπει να επεταχυνθούν και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα τελευταία μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αυτές οι δραστηριότητες στην αρχή της νέας περίοδου ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαρύνουν την ημερήσια διάταξη, ε, πρέπει όμως να πετύχουμε και ε, με ενθαρρύνει και η ταχύτητα με την οποία τα θεσμικά όργανα κατέληξαν σε συμφωνία για τις προηγούμενες προτάσεις για το Brexit. Η Προεδρία του Συμβουλίου με την συνεργασία σας είναι διατεθειμένη να διευκολύνει την υιοθέτηση των έκτακτων μέτρων τα οποία θα χρειαστούν. Θα εξαρτηθεί το σημείο εκκίνησης για τις επόμενες σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο για το από το αν θα αποχωρήσει με τακτικό ή μη τρόπο θα πρέπει να διασώσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να τιμήσει τις υποχρεώσεις του που προέρχονται από την ιδιότητά του ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουμε φυσικά την σταθερότητα και την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς όπως και τη σταθερότητα στην Ιρλανδία. Η αβεβαιότητα αυτή και οι εντάσεις οι οποίες ε, προκαλούνται ε, θέτουν σε δοκιμασία την ενότητά μας. Είναι απαραίτητο συνεπώς λοιπόν να αρνηθούμε την πρόκληση των διμερών συμφωνιών σε τομεακές ε, περιπτώσεις και δεύτερον να υιοθετηθούν τα έκτακτα αυτά μέτρα το ταχύτερο δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να πω ότι και στο δικό σας ψήφισμα προτείνονται ε, θέματα τα οποία ε, είναι θα έλεγα ταυτόσημα με τις προτεραιότητες του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει για την προσοχή σας και περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ την Υπουργό και θα δώσω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο κύριο Γιούγκερ τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του στην αίθουσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να πάρω το λόγο ενώπιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μιλήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα βασίστηκε στην συνεργασία ε, και στις καλές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό σχετίζεται και με τα όσα πετύχαμε μαζί για το θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ξέρω πως εσείς είστε πάντα ανοιχτοί και πάντα κάνετε τη δουλειά σας. Ο Μισελ Μπαρνιέ και εγώ γευματίσαμε τη Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό κύριο Τζόνσον δεν θα σας εκπλήξω το γεγονό πως ο Πρωθυπουργό μας είπε ε, πως το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να επιθυμεί συμφωνία, αλλά πως θα φύγει οπωσδήποτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 31 Οκτωβρίου με ή χωρί συμφωνία. Αυτό δεν έχει μεταβληθεί. Τι σημαίνει τούτο. Πως ο κίνδυνος του no deal παραμένει πολύ υπαρκτός. είναι η οπαδή μου, το fan club. Μη σα ε, εντυπωσιάζει που με χειροκροτούν. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι πως υπάρχει υπαρκτός κίνδυνο που είναι επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δική μας επιλογή τούτο που δεν θα είναι ποτέ. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ στα όσα μπορούμε να κάνουμε για να βρούμε στο μέλλον μια συμφωνία, μια συμφωνία την οποία θεωρώ ευκταία και πάντα βιώσιμη. Πρέπει να με χειροκροτήσετε. Στρεφόμενος προς τα έδρανα. Δεν θα σε, σας εκπλήξει καθόλου πως το βασικό θέμα είναι το δίκτυ ασφαλείας, το backstop, γιατί νομίζω πως όλοι το έχετε ακουστά. Αλλά δεν θυμόσαστε όλοι τους λόγους για τους οποίους συμφωνήθηκε ε, μεταξύ των 27 κρατών μελών και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το backstop είναι μια λύση ε, λειτουργική για ένα πρακτικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί το Brexit ε, για το νησί της Ιρλανδίας. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα είχε εμφανιστεί αν δεν είχε αποφασίσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει. Το backstop προσπαθεί να εξυπηρετήσει τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να μην υπάρχει φυσικό σύνορο στο νησί της Ιρλανδίας, να διατηρήσει την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς και κυρίως τη θέση της Ιρλανδίας σε αυτή την ενιαία αγορά και επίσης να προστατεύσει την νησιωτική αυτή οικονομία ολόκληρου του νησιού και τις σχέσεις βορρά και νότου στο νησί. Γιατί ξέρετε όπως έχουμε στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, τοποθετήσει κάποιες αρχές τις οποίες θα πρέπει πάντα να σεβόμαστε. Και είχε συμφωνηθεί, εγώ πάντα είπα πως μπορεί το backstop να έχει κάποια άλλη μορφή, αλλά αυτούς τους τρεις στόχους πρέπει οπωσδήποτε να τους πετύχουμε. Και γι' αυτό είπα στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να μας κάνει πρακτικές, γραπτές και λειτουργικές προτάσεις για κάτι άλλο που θα επέτρεπε να πετύχουμε αυτούς ακριβούς τους στόχους. Όσο δεν είναι στο τραπέζι τέτοια πρόταση, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε ένα στα μάτια και να πούμε πως έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος. Αυτό το οποίο είπα γιατί γράφουν πολλά στο βρετανικό τύπο, αυτό που είπα ήταν πως ήταν επικοδομητικές οι συζητήσεις μας και σε κάποιο βαθμό θετικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εργαστεί κάθε μέρα πρωί βράδυ. Εντάξει, θα κάνουμε και κάποιες ψηλοδιακοπές, αλλά θέλουμε να βρούμε κάποιες τεχνικές και πολιτικές λύσεις. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος πως θα το πετύχουμε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας, αλλά είμαι σίγουρος πως θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Ζήτησα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό να μας διευκρινίσει ποιες είναι οι εναλλακτικέ διαφθετήσεις τις οποίες θα μπορούσε να δεχτεί και πρότεινα να πολιτικοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτοντας το φίλο Μισελ Μπαρνιέ και τον ομόλογό του στη Βρετανία να αναλάβουν οι ίδιοι τα ενία στις διαπραγματεύσεις μια και ε, υπάρχουν κάποια θέματα που ξεπέρνουν το τεχνικό. Να σας πω πως οι 27 αναγνώρισαν πως θα ήταν ε, λάθος όλη μας την ενέργεια να την επικεντρώσουμε στο Brexit. Είπαμε πως θέλουμε μια πιο βαθιά ένωση και θα πρέπει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας. Αυτά τα είπαμε το 2016. και δύο χρόνια μετά μίλησα στο Κοινοβούλιο και περιέγραψα την κατάσταση της Ένωσης και σας είπα ποιες είναι οι προτάσεις μου. Ο λόγος αυτός επικροτήθηκε από όλους τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην Πρατισλάβα που είχαμε μαζευτεί και πρέπει να σας πω τα εξής. Και όταν λέω 27, εννοώ πως οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για δυόμιση χρόνια διαπραγματεύονται με το Ενωμένο Βασίλειο για να προσπαθούμε τις σχέσεις μας να τις οργανώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε μεγάλη ενότητα και Ήτανε απόλυτα αφοσιωμένη στο στόχο αυτό για να στηρίξει τα κράτη-μέλη τα οποία ε, βρίσκονται ε, σε μεγαλύτερη δυσκολία από το θέμα αυτό. Και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε τις επόμενες εβδομάδες και είμαι σίγουρος πως θα ε, συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να καθοδηγούμε και τα πάντα και εδώ στο άμεσο και μακρινό μέλλον. Ευχαριστώ τον κύριο στον κύριο διαπραγματευτή τώρα, τον κύριο Μπαρνιέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε μετά τον Πρόεδρο Γιούνκερ, συμπληρώνοντας αυτά που πολύ ξεκάθαρα μας είπε, να επανέλθω με μια σύντομη παρέμβαση και να μιλήσω για τα δύο βασικά σημεία της τωρινής μας συζήτησης με τους Βρετανούς το θέμα της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και το θέμα της μελλοντική σχέσης, που είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική, διότι θα πρέπει με ένα διαφορετικό τρόπο να ξαναχτίσουμε μια εταιρική σχέση με αυτές τις δύο φίλες και γείτονες ε, σχέσεις, γιατί, ε, γείτονες χώρες, γιατί θα παραμείνουν φίλες και γείτονες χώρες αυτές. Το θέμα το οποίο συζητάμε με τον, ε, πρόεδρο, με τον Πρωθυπουργό συγγνώμη, Τζόνσον είναι το backstop, το δίκτυο ασφαλεία ε, και ενδεχομένω η αντικατάστασή του. Ξέρετε ότι συμφωνήσαμε το Νοέμβριο του 2018, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, για αυτό το μηχανισμό ασφαλεία. Συμφωνήθηκε λοιπόν από του 28 αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων με ισχυρή υποστήριξη από το δικό σα κοινοβούλιο και γιατί είναι τόσο θεμελιώδες αυτό το θέμα για όλους μας. Πολύ απλά και ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα, διότι στην Ιρλανδία δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα το Brexit. Στην Ιρλανδία υπάρχουν οι περισσότεροι κίνδυνοι λόγω του Brexit. Είναι το μόνο σημείο στο οποίο έχει χερσαία σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει μια ιδιάζουσα πολιτική κατάσταση που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι συνδέεται ε, η ιστορία που μερικές φορές είχε και τραγικά συμβάντα και τώρα με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν εγγυηθεί αυτή την ε, σταθερή πολιτική κατάσταση οι λόγοι για τους οποίους το συζητάμε δεν είναι ιδεολογικοί, όπως είπε ο, κύριος, ο πρόεδρος Γιούγκα, είναι απόλυτα ρεαλιστικοί. Μέσω του μηχανισμού ασφαλείας, που αποκαλούμε backstop, θέλουμε να έχουμε μία διασφάλιση που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις τις τρεις απαιτήσει που υπενθύμησε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν θέλουμε να ξαναέχουμε φυσικό σύνορο στην Ιρλανδία. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε όλες τις διαστάσεις της. Πρέπει να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς, ε, της δικής μας ενιαίας αγοράς και θέλουμε να διατηρήσουμε την οικονομία σε ολόκληρο το νησί, συνεργασία μεταξύ Βορρά και Νότου, εφαρμόζοντας την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Και υπενθυμίζω ότι η διαδικασία χαρτογράφησης που κάναμε με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε πόσο αυτή η συνεργασία Βορρά-Νότου υποστηρίζεται και πρέπει να υποστηρίζεται από τους πολιτικούς και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο εξ αρχής συνέβαινε. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μας εξήγησε και αυτή τη βδομάδα στο Λουξεμβούργο τι δεν της αρέσει στο backstop. Αλλά δεν αρκεί να μας εξηγούν γιατί θα έπρεπε να καταργήσουμε το backstop. Εμείς από την πλευρά μας πολύ απλά και με μεγάλη σοβαρότητα χρειαζόμαστε λύσεις που να είναι νομικά λειτουργικές στη συμφωνία αποχώρησης για να μπορεί όλα αυτά τα προβλήματα και κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα να αποτρέπονται, να αποτρέπονται όλοι οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τον Brexit. Και αυτός είναι ο στόχος που θέσαμε σαφώς με την κυβέρνηση της Τερίζα Μέη. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα θα σας φέρω, το οποίο το γνωρίζω αρκετά καλά, διότι ήμουν υπουργό Γεωργίας και Αλίας πριν από λίγα χρόνια. Όλα τα ζώντα ζώα και όλα τα προϊόντα, όλα τα τρόφιμα συγκεκριμένα που φτάνουν στη Βόρεια Ιρλανδία με προέλευση τη Μεγάλη Βρετανία έχουν όχι μόνο στην ίσο της Ιρλανδίας, ε, μπαίνουν, μπαίνουν όχι μόνο στην ίσο ε, της Ιρλανδίας, αλλά και στην αγορά της Πολωνίας, της Δανίας, άμεσα, με μηχανικό τρόπο, μπαίνουν στην ε, νέα αγορά. Και πρέπει να ασκούμε ένα έλεγχο, γιατί οφείλουμε να προστατεύουμε τους καταναλωτές, να προστατεύουμε όλους ε, τους ευρισκόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ε, ζωικές ε, νόσους και θέλουμε να προστατεύουμε και τους καταναλωτές της Βορείου Ιρλανδίας και ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου και ολόκληρης της νήσου της Ιρλανδίας. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένες εγγύησεις τις οποίες χρειάζονται όλοι οι πολίτες στην ίσο της Ιρλανδίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα, για την ε, καθημερινή ε, οικονομική ζωή και για την υγεία των καταναλωτών των 27 κρατών μελών, για την προστασία των εθνικών προϋπολογισμών, γιατί οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ε, ενιαίας αγοράς σε αυτό αποσκοπούν. Ακούσαμε και τις παρατηρήσεις του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ε, δημοκρατικό ή μη δημοκρατικό χαρακτήρα του backstop. Η ίδια η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει ε, να εξασφαλίσει στη Συμφωνία Αποχώρησης το δημοκρατικό χαρακτήρα. Στη Συμφωνία Αποχώρησης έχουμε ήδη πολλές διατάξεις, ιδίως για το πώς θα υπάρχουν διάφορες επιτροπές και θεσμοί για την εφαρμογή του backstop εάν χρειαστεί να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή. Και για αυτό το ερώτημα, όπως και για όλα τα άλλα, είπα, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ... ότι είμαστε διαθέσιμοι, θα ακούσουμε τους Βρετανούς και θα δουλεύουμε μέρα νύχτα εφόσον οι προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μας παρουσιάσουν κάποια εξέλιξη. Ένα άλλο θέμα κλειδί και θα κλείσω με αυτό το βασικό θέμα, είναι το θέμα της κοινή μας φιλοδοξίας για τις μελλοντικέ σχέσεις. Την στρατηγική εταιρική σχέση, όπως την αποκαλέσαμε, την οποία πρέπει να χτίσουμε ή να ξαναδημιουργήσουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Και αυτό είναι το αντικείμενο του δεύτερου εγγράφου, παράλληλα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, έχουμε και την πολιτική διακήρυξη που συμφωνήθηκε μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο το Νοέμβριο του 2018 και που ανοίγει το δρόμο σε αυτή την ευρεία εταιρική σχέση για οικονομική συνεργασία, τομεακή συνεργασία, δικαστική, αστυνομική συνεργασία, συνεργασία σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Το οικονομικό κομμάτι, αυτή η εταιρική σχέση παίρνει τη μορφή μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Αλλά στο τωρινό κείμενο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φιλοδοξίας. Εμείς έχουμε τη βούληση να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι σε αυτή την εταιρική σχέση και την οικονομική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Παραδείγματο χάρη μέσω μιας τελωνιακής ένωσης. Αυτές οι οικονομικές σχέσεις θα πρέπει βεβαίως να συνοδεύονται από εγγύησεις για ε, ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Αναγνωρίζω ότι οι δίκαιε συνθήκε ανταγωνισμού είναι ένα όρο αρκετά τεχνικό. Πίσω από αυτόν τον όρο υπάρχουν και ανθρώπινε, κοινωνικέ και εδαφικέ ε, πραγματικότητε. Και αυτό είναι μια επιλογή που θα πρέπει να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ του ορθού επίπεδου ρύθμιση και ε, των οικονομικών συνθήκων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να επανέλθει από αυτού, θέλει να επανέλθει επί των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Τερίζα Μέη στον τομέα των δίκαιων συνθήκων ανταγωνισμού. Με μια μεγάλη χώρα τόσο γειτονική και τόσο σημαντική όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που το ίμιση του εμπορίου του το υλοποιεί με εμά, με την ενιαία αγορά, πρέπει να έχουμε και φιλόδοξες βλέψεις, αλλά και μία βάση για κοινούς κανόνες του παιχνιδιού. Το λέω λοιπόν για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα προς όλους, ότι το επίπεδο φιλοδοξίας για μια μελλοντική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που πρέπει να διαπραγματευτούμε και να συνάψουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας θα εξαρτηθεί σαφώς από τις εγγυήσει που θα έχουμε βάλει επί χάρτου για κοινωνικά, περιβαλλοντικά, θέματα ανταγωνισμού και θέματα δημοσίου χρέους. Ήθελα να μιλήσω για αυτά τα δύο θέματα τα οποία συζητούνται τώρα με την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον χωρίς να χάνουμε βέβαια τη συνολική εικόνα. Και κλείνοντας θέλω να υπενθυμίσω γιατί θελήσαμε εξ αρχής να έχουμε μία συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πολύ προτιμότερη από την ε, απουσία συμφωνίας. Και όταν μιλάμε για απουσία συμφωνία, για αποχώρηση χωρί συμφωνία, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τι συνέπειε για το Ηνωμένο Βασίλειο καταρχήν, αλλά και για μα. Τι συνέπειε τη απουσία μια συμφωνία. Τη συμφωνία αυτή τη χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των 4,5 εκατομμυρίων πολιτών και πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολείπων κρατών μελών σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους, να εξασφαλίσουμε το μέλλον των ευρωπαϊκών έργων και γι' αυτό μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήσαμε ότι ό,τι έχει συμφωνηθεί από τους 28 θα πληρώνεται μέχρι τέλους από τους 28. Θέλουμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητα στην Ιρλανδία, στην ίσο της Ιρλανδίας και θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες απαραίτητης εμπιστοσύνης για να χτίσουμε τη μελλοντική μας σχέση όπως ε, διαγράφεται στην πολιτική διακήρυξη. Εάν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία, Θέλω να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι όλα αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Όλα αυτά στη Συμφωνία Αποχώρησης τα έχουμε ρυθμίσει. Αλλά παραμένουν ως θέματα τι θα γίνει με τους πολίτες, η ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία η ενιαία αγορά, όλα αυτά τα θέματα του προπολογισμού, όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν και θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ των προτέρων για μια μελλοντική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συνέπειε του Brexit δεν είναι θεωρητικέ και πολλέ φορέ εδώ στο ημικύκλιο σα έχω πει ότι είναι αμέτρητε και συχνά τι υποτιμούμε όσον αφορά το ανθρώπινο και κοινωνικό πεδίο, όσον αφορά το οικονομικό, το δικαστικό, το τεχνικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικέ οι συνέπειε. Και το υπενθυμίζετε κι εσείς ε, άλλη μια φορά σήμερα στο ψήφισμά σας. Περίπου τρία χρόνια μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα, δεν θέλουμε να προσποιούμεθα ότι διαπραγματευόμαστε. Έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε αυτές τις διαδικασίες με αποφασιστικότητα, με ειλικρίνεια και θα συνεχίσουμε με συνεχείς διαβουλεύσεις με κάθε διαφάνεια με τις κυβερνήσεις ε, των ε, κρατών μελών και ευχαριστώ την Προεδρία. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τις προσπάθειές σας και θα συνεχίσουμε και με την ε, ομάδα καθοδήγησης για τον Brexit και την ομάδα συντονισμού για τον Brexit με το κοινοβουλίο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή θα παραμείνει η στάση μας σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες και σύνθετες διαδικασίες. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ε, μετά τον κύριο Μπαρνιέ θα ακούσουμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές οι μπλε κάρτες. Ο κύριος Βέμπερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Μπαρνιέ, Τρία χρόνια μετά το δημοψήφισμα οι οπαδοί του Brexit λένε ότι τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόκειται να συνεχίσει να λειτουργεί μετά την αποχώρησή μας. Τρία χρόνια μετά όμως εξακολουθούμε να είμαστε εδώ. Δυστυχώς η Βρετανία δεν φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα αλλά θέλει να φύγει. Οι επιχειρήσεις όμως θέλουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1 τρίτο των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρούν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Ε, κατά τη διάρκεια των εκλογών ήταν ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα το οποίο έδειξε στους Ευρωπαίους ότι δεν πρέπει να αμφισβητείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πείσαμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενδιαφερθούν και να προστατεύσουν την Ευρώπη. Ο κύριος Μπαρνιέ, ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Τζόνσον πριν λίγες μέρες είχαν την δυνατότητα να διευκρινίσουν τα πράγματα και να συζητήσουν νέες προτάσεις. Εμείς συζητάμε την κατάσταση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι την Κάτω Βούλη λένε ότι το Westminster θα αναλάβει πια την τύχη της χώρας, έλεγε ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και γι' αυτό έκλεισε την κάτω βουλή προσωρινά. Ακύρωσε τη λειτουργία της. Κυρίε και κύριοι, σκέφτομαι ότι η εκπροσώπηση του λαού μέσω του ε, Πρωθυπουργού θα πρέπει να εκπροσωπεί πραγματικά το λαό. Το 51% αποτελεί πλειοψηφία και πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά 51% ως έκβαση του δημοψηφίσματος δεν αποτελεί το σύνολο του λαού. Το σύνολο του λαού εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Εκεί εκφράζονται ε, ε, οι απόψεις του λαού δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι παρά τη θέληση και εναντίον της θέλησης του Κοινοβουλίου. Αυτό ε, θέτει σε κίνδυνο την κοινωνία μας, γιατί ε, η ηγετική στάση σημαίνει όχι διχασμό, αλλά η ηγετική στάση σημαίνει συνένωση του λαού. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι σαφές ότι θα υποστηρίξουμε το σημερινό ψήφισμα και ευχαριστώ τον Μισελ Μπάχνια για τη δουλειά του και ευχαριστώ και τον ε, Γκίφερ Χόφστατ και όλου όσου συμμετέχουν στην ομάδα συντονισμού για το Brexit. Δείχνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενωμένο προχωρεί σε αυτή τη συζήτηση και μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλά καλά επιχειρήματα σε αυτά που αναφέρονται και θα πρέπει σε όλες τις προτάσεις που συζητούνται τώρα να είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να επιτρέψει δίπλα στην πόρτα μας να υπάρχει κάποιο dumping παρά τα πρότυπα τα οποία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το αναφέρω ως προειδοποίηση. Έχει γίνει πλέον ε, απρόβλεπτο το Brexit και γι' αυτό θα πρέπει ε, ε, να είμαστε σε επαγρύπνηση. Θα πρέπει οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες έχει το λόγο. Ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα ήταν κακή είδηση για όλους μας, αλλά κυρίως θα ήταν καταστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με τη δική μας γνώμη. Η πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσης Yellowhammer από την Βρετανική κυβέρνηση προειδοποιεί για τα χειρότερα σενάρια ενός Brexit και καταρρύπτει αυτή την ουτοπία την οποία έχει χτίσει ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος θεωρεί πως ε, η τιμή του ηλεκτρικού η διέλευση της μάχης, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, όλα αυτά θα πλήξουν τους πιο αδύναμους οικονομικά και βέβαια η ε, αβέβαιη θέση των Βρετανών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να αλλάξω τη στάση συγκεκριμένων ευρωβουλευτών για το θέμα αυτό. Το μόνο που ζητώ είναι σεβασμό. Δεν είμαι αφελής, δεν ζητώ να σεβαστείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε χρόνια που δεν μας σέβεστε. Να σεβαστείτε το λαό τον οποίο λέτε πως εκπροσωπείτε. Γιατί τα γέλια σας θα γίνουν αβεβαιότητα, δάκρυα και φόβοι για εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν το τι θα βγει από τη δική μας συζήτηση. Και να σας πω πως αυτό το πλαίσιο οι βασικές προευρωπαϊκές δυνάμεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του ψηφίσματος δείχνουμε τη στεναρή μας στήριξη για μια επέκταση του άρθρου 50 για να αποφύγουμε το καταστροφικό σενάριο που είναι η μη συμφωνία αν το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται χρόνο για να κάνει εκλογές ή καινούριο δημοψήφισμα. Θα μπορείτε να βασιστείτε στη δική μας στήριξη. Και ξέρετε ποιος δημιούργησε το χάος αυτό. Θα σας πω τον όνομα του υπευθύνου για το χάος. Μπόρις Τζόνσον. Και λέγαν παλιά πως το όνομα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ε, και το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνας. Ε, ακούσατε τα όσα είπε για τον Τσέρτσιλ και για το τι σημαίνει Βρετανός ηγέτης. Νομίζω πως η τύχη επιφυλάσσει ε, για τον Μπόρις Τζόνσον να είναι αυτός που θα επιβλέψει ε, την καταστροφή του συνδέσμου που είχε δημιουργήσει ο μεγάλος αυτός πολιτικός μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης. Εδώ οι σοσιαλιστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτούμε από τον Μπόρις Τζόνσον και από την κυβέρνησή του να εξασφαλίσουν τα κεκτημένα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στην στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ουσιαστικό θέμα και μας ανησυχούν πάρα πολύ οι διάφορες δηλώσεις που έχει κάνει η Υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας για τη λήξη της ελεύθερης κυκλοφορίας από τις 31 Οκτωβρίου και μετά. Οι πολίτες δεν πρέπει ποτέ να πληρώσουν το αντίτιμο για τα λάθη που κάνουν οι ηγέτες τους. Αυτό είναι σαφές. Και η δική μας προτεραιότητα είναι η συντεταγμένη αποχώρηση. Και γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε το εργαλείο της συμφωνίας, γιατί έτσι δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ του ΕΙΡΕ και της Βορείου Ιρλανδίας, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα ε, ε, των Ευρωπαίων πολιτών Έχουμε διαπραγμάτευτη την ακαιρεότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Είναι ιστορικό το λάθος και εμείς θα στηρίξουμε τον Βρετανικό λαό αν αποφάσει να αντιστρέψει αυτή την απόφαση. Και καλά θα έκανε να θυμάται ο Βρετανός Πρωθυπουργό τα όσα είχε πει ε, στις Βρυξέλλες ο Winston Churchill που ήταν ο ήρωας παιδική τους ε, ηλικίας. 20 Νοεμβρίου του 1945 είχε πάει στο Βελγικό Κοινοβούλιο και είχε πει δεν βλέπω γιατί δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Και με τον τρόπο αυτό θα δυναμώσουμε τον, ε, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θα ζήσουν οι λαοί μας μαζί σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει διακόψει τη λειτουργία του, αλλά με τη συζήτηση την οποία κάνουμε δείχνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σταματήσει τη λειτουργία της. Είναι καταπληκτικό το ότι το κόμμα Brexit και ο κύριος Φαράζ κάνουν τέτοια φασαρία. Δεν μπορούν να το κάνουν στο δικό τους κοινοβούλιο τη φασαρία αυτή και την κάνουν εδώ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν εκλεγεί στο Westminster. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι ευρωσκεπτικιστές, ε, λέτε συνέχεια πράγματα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέτε ότι είναι αντιδημοκρατική και σε λίγα δευτερόλεπτα το ίδιο θα μας πείτε για μια ακόμη φορά. Να πω όμως ότι ο Γιούνκερ και ο Τούσκ μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούν να διατάξουν να σταματήσει η λειτουργία αυτού του κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε γελίες συγκρίσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προσπαθήστε να το κάνετε και στο Westminster και όχι μόνο στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Η ελπίδα την οποία έχω είναι ότι το ψήφισμα και ε, η ψηφοφορία θα δείξει την ενότητα που έχουμε σε σχέση με τον Brexit. Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο και τα 27 κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν συζητήσεις γύρω από αυτό. Το Brexit είναι κάτι το κακό, είναι μια κακή ιδέα, αλλά έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ε, επανένωσε τους Ευρωπαίους και το ευρωπαϊκό σχέδιο αν θέλετε μετά το Brexit έχει γίνει πολύ πιο δημοφιλές από ό,τι ήταν πριν το Brexit. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα των λαών κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών ήταν σημαντικά. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Ε, προστατεύουμε την Ευρώπη. Δεν φεύγουμε από την Ευρώπη. Και αυτό ίσχυσε και ε, στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά ε, και στις ευρωεκλογέ στη Μεγάλη Βρετανία. 40 Βρετανοί ευρωβουλευτές είναι οι λεγόμενοι remainers, είναι υπέρ της παραμονής. Αυτό είναι, αυτά είναι τα πράγματα σήμερα. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και εμείς βάζουμε τρεις προϋποθέσεις γι' αυτό και θα ήθελα να υπενθυμίσω Πρώτον, ε, διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών και των Βετανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε πετύχει στην παρούσα στιγμή. Καθημερινά στον Βρετανικό τύπο ακούγονται προτάσεις και περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν δεκαετίες ολόκληρες στη Μεγάλη Βρετανία και δεν έχουν ε, ξεκάθαρο καθεστώς παραμονής. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται ένας πολύ σημαντικός τρόπος αλλαγής της διαχείρισης αυτού του τμήματος της Συμφωνίας Αποχώρησης. Δεν θέλουμε μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση όπως η σημερινή. Αυτό που περιμένουμε από, το Βρετανικό, από τη Βρετανική πλευρά είναι η αυτόματη αδειοδότηση παραμονής των Ευρωπαίων πολιτών. Γνωρίζω ότι ο κύριος Μπάρις Τζόνσον συγκρίνει τον εαυτό του με διάφορα κινούμενα σκίτσα. Και γι' αυτό σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών, αντί να παίζει τον οργισμένο Χάλκ, ας επιλέξει έναν άλλο βουλευτή, την κυρία Φάιερ από τον κινηματογράφο, δηλαδή την Νταντά που προστατεύει τα παιδιά. Θα επανέλθω λοιπόν τώρα να, στο λεγόμενο σύνορα στην Ιρλανδία. Backstop αν θέλετε ή κάτι, κάποια άλλη λέξη. Θέλετε να χρησιμοποιούμε τον όρο δίκτυα ασφαλείας. Γιατί όχι, ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Απαιτείται ένα τέτοιο δίκτυο ασφαλείας και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Ο βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε ανάγκη είναι η βία να μην επιστρέψει στο νησί της Ιρλανδίας. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Και πρέπει να σας πω ότι βρίσκω εντελώς ανεύθυνο από πλευρά ορισμένων βουλευτών και σκληρών συντηρητικών που δεν δέχονται την πρόταση στην οποία είχαν καταλήξει παλιότερα. Τη στιγμή που συζητάμε, και ερωτώ τον κύριο Γιούνκερ και τον κύριο Μπαρνιέ αν μπορούν να το επιβεβαιώσουν, δεν έχει υπάρξει καμία νομικά δεσμευτική και εφικτή και πρακτική πρόταση από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το backstop λοιπόν, όπως το περιγράφει ε, ο αγγλικός τύπος σήμερα για τον περιορισμό του backstop στα γεωργικά προϊόντα. Δεν αρκεί αυτό, δεν αντιπροσωπεύουν παρά το 30% των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και το θέμα της απόφασης την οποία θα λάβει το Stormont δεν έχει άμεση σχέση με το backstop γιατί θα είναι ένα μόνιμο μέσο εκβιασμού της, ενώ με το Stormont την τοπική βουλή στη Βόρεια Ιρλανδία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στην Ιρλανδία και στον υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια τελευταία παρατήρηση τώρα για τις μελλοντικέ σχέσεις. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε ένα νέο κοινοβούλιο. Άνω του 60% των μελών είναι νέοι βουλευτέ. Πρέπει να το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά. Το κοινοβούλιο αυτό δεν θα δεχθεί ποτέ μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Μεγάλη Βετανία θα έχει όλα τα πλεονεκτήματα τη ελεύθερη αγορά, μηδενικού δασμού και δεν θα υπακούει του κανόνε στον τομέα τη οικολογία και τη κοινωνική πολιτική στο μέλλον. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πολλοί Βρετανοί λένε έτσι κι αλλιώς οι Ευρωπαίοι στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα υποχωρήσουν. Όχι, δεν είμαστε τόσο ανόητοι και αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα δολοφονήσουμε τις επιχειρήσεις μας, θα τις υπερασπιστούμε. Θα υπερασπιστούμε τις οικονομίες μας, θα υπερασπιστούμε την ενιαία μας αγορά και δεν θα δεχθούμε ποτέ αυτό το οποίο πολλοί ονομάζουν η Σιγκαπούρη της Βόρειας Θάλασσας. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Τέλος. Ξέρετε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε το Brexit. Ήταν μια απόπειρα του Κάμερον να καλύψει τις διαφωνίες που υπήρχαν στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος. Οι συνέπειες είναι τεράστιες διαιρέσεις στην ίδια τη Βρετανική κοινωνία. Εμείς ε, δεν θα επιτρέψουμε το Brexit αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ κύριε Βερχώστα. Το κύριος Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν επιλέξαμε το Brexit. Όμως σεβόμαστε την επιλογή που έχει κάνει μια πλειοψηφία των Βρετανών ε, και γι' αυτό θα διαπραγματευτούμε μία συμφωνία η οποία θα επιτρέψει αυτή τη ε, διαίρεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμε θα ιδιαίτερα. Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απελευθερώνει το Ηνωμένο Βασίλειο από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει ε, αποκτήσει εδώ και 45 χρόνια που είναι νομικά δεσμευτικές ε, για παράδειγμα αυτές της ε, συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής ε, που έφερε σε, ε, να κλείσει μια σύραξη που κόστησε 3.000 ζωές. Ο, Ηνωμένος, ο, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και πολλοί πολιτικοί μοιάζουν να αγνοούν το γεγονός πως έχουν αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις. Γιατί η θέση που εκφράζει ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι, και το λέω συνοπτικά, να λέει στους Ευρωπαίους σας λέω να ανοίξετε ένα διάδρομο 500 χιλιόμετρα στην ενιαία αγορά και εμείς θα κάνουμε dumping κοινωνικό, φορολογικό και επιβαλλοντολογικό όσο επιθυμούμε. Μα αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και αυτό δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε 27 αρχηγούς κρατών ε, μελών και δεν θα δημιουργήσει την εμπιστοσύνη και τη σχέση εμπιστοσύνης που χρειαζόμαστε για να ε, διαπραγματευτούμε μια συμφωνία. Και δυστυχώς είναι ακόμα στην καυτή επικαιρότητα η δυνατότητα της αποχώρησης χωρίς συμφωνία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να βάλουμε στην άκρη. Και ρωτώ το Ηνωμένο Βασίλειο, τι φαντάζεστε πως θα συμβεί αν κάναμε κάτι αντίστοιχο εμείς 27 με την Κίνα. Τι σημαίνει αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Τι σημαίνει το να βλάψεις την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς 27 κρατών μελών. Τι θα επιλέξεις. Θα επιλέξεις το μη χείρον βέλτιστον. Αυτό λοιπόν που ζητώ είναι το εξής. Να απευθυνθούμε στα εκατομμύρια ευρωτενού που γνωρίζουν πού είναι το συμφέρον της χώρας τους, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λέω εδώ, σαφέστατα, αν το Ηνωμένο Βασίλειο είτε μέσω Πρωθυπουργού ή με οποιαδήποτε άλλη αρχή ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία επέκταση της προθεσμίας για το άρθρο 50, εμείς πρέπει να δεχτούμε αυτό το αίτημα. Όσο υπάρχει η δυνατότητα η λογική να πρετανεύσει, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο, ο πρόεδρος Τζάνι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ εντυπωσιάζομαι πολλές φορές από την περιφρόνηση εναντίον της δημοκρατίας δίνουμε μαθήματα δημοκρατίας σε μια από τις παλαιότερες δημοκρατίες του κόσμου, σε ένα από τα πιο παλιά κοινοβούλια του κόσμου. Όταν αυτό το κοινοβούλιο έχει επιδείξει για πάρα πολλά χρόνια ότι πραγματικά αποστρέφεται τις δημοκρατικές αρχές, αποκλείει τις μειονότητες από την εκπροσώπηση και ακολουθεί διαδικασίες αποφάσεων, λήψης αποφάσεων που δεν ελέγχονται από το Κοινοβούλιο αλλά από γραφειοκράτες ανεξέλεγκτους. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό περιλαμβάνεται και στην ουσία των ψηφι, του των θέσεων του ψηφίσματος ε, το οποίο ε, θα υπεψηφίσει από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση της, του δημοκρατικού καθήκοντος όπως ένα δημοψήφισμα είναι κάτι το θλιβερό και κάνετε μαθήματα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ε, και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η αποστροφή που έχετε για τη δημοκρατία δεν έχει σχέση μόνο με το Brexit, αλλά στην πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία τα ευρωπαϊκά όργανα περιφρονούν τις αποφάσεις των πολιτών. Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Έλληνες οι οποίοι είπαν όχι ε, στις παρεμβάσεις των Βεξελών, αλλά ξέρουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν μετά να δεν ανησυχώ εγώ για το κλείσιμο της Βρετανικής Βουλής. Είναι μια πρακτική η οποία προβλέπεται από το Βρετανικό Σύνταγμα. Εμένα με απασχολεί η αποστροφή του Κοινοβουλίου για τις εκλογικές διαδικασίες και τα δημοψηφίσματα. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται ελεύθερα από τους λαούς που δεν αρέσουν αυτές οι αποφάσεις στα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου θα πρέπει και με ανορθόδοξους τρόπους να αλλάξουν. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι το πραγματικό θέμα του Brexit είναι ο φόβος τον οποίο έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα, ο φόβος ότι κάποιος άλλος διαλέγει έναν άλλο δρόμο, ο φόβος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδείξει ότι το ευρωπαϊκό όργανο δεν είναι τέλειο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η μοναδική λύση και ότι μπορεί κάποιος να ακολουθήσει μια διαφορετική οδό και να πάει καλύτερα. Αυτή είναι η ελεύθερη επιλογή των Βρετανών συνοδέλφων και πρέπει να τους σεβαστούμε. Το να θελήσουμε να συγκρουστούμε και να θελήσουμε να τιμωρήσουμε τους πολίτες του Ενωμένου Βασιλείου γιατί αποφάσισαν να ακολουθήσουν μία άλλη οδό δεν τιμά το δικό σας ίδιο το πολιτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είδα από πλευρά των μελών του Κοινοβουλίου να εξετάζουν πραγματικά το τι λέει η συνείδησή τους, το αν προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ένα κράτος μέλος αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ένα κράτος μέλος αποφάσισε να πει ως εδώ και εγώ βλέπω το τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό που με ανησυχεί επίσης είναι η μεγάλη θεσμική και πολιτική κρίση η οποία χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες μέλη, προβλήματα και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που ε, μπόρεσαν με οριακό τρόπο να επιλέξουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς λοιπόν δεν πρέπει να εμποδίζετε άλλους να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο, αλλά καλύτερα να σκεφτείτε τα προβλήματα τα οποία εσείς ήδη έχετε, γιατί αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα μέλλον. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος Φανόρντεν έχει το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστώ τον Ζων Κλοντ Γιούνκερ και τον Μισελ Μπαγνιέ για τις ε, πολύ χρήσιμες ε, και γενικές παρατηρήσεις του σήμερα το πρωί το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θέλει μια συμφωνία, όχι οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά μια που να είναι αποδεκτή και από το λαό. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε αυτή τη συμφωνία σύντομα για να μπορέσουμε να φύγουμε στι 31 Οκτωβρίου. Επρόκειτο να φύγουμε το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τώρα στι 31 Οκτωβρίου. Ποιο είναι ο λόγο για περαιτέρω καθυστέρηση. Κάποιοι από εσά μπορεί να πιστεύετε ότι αν ε, συνεχίσουμε με αυτή την καθυστέρηση, μπορεί να έχουμε αλλαγή καθεστώτο ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλαγή γνώμη. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτη ψευδέστηση. Οι μελλοντικέ σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται σε σχέσεις ε, φιλίας ε, και καλής γειτονίας και όχι σε θυμό και εμνηση Χρειάζεται καλή θέληση και ευελιξία για να επιταχύνουμε τις προσπάθειες και από τις δύο πλευρές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα δεν είναι εφικτό και τα πάντα είναι εφικτά. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφέ για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ευπρόσδεκτοι και θα προστατευτούν τα δικαιώματά του. Και πάνω από ένα εκατομμύριο ετούντε ήδη έχουν πάρει ε, άδεια παραμονή και έχουν χρόνο και όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν αίτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια εξίσου γενναιόδορη προσέγγιση προ του ε, πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόβλημα που παραμένει είναι βέβαια τα σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Κανείς δεν θέλει να αμφισβητήσει την ειρηνευτική συμφωνία. Ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν παραμένουμε πιστοί στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή η συμφωνία δεν αναφέρει τα σύνορα. Βασίζεται όμως ε, στην ε, εκτίμηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, των δύο παραδόσεων στην ίσο της Ιρλανδίας. Και μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι στην Βόρεια Ιρλανδία είναι ενωτικοί, είναι υπερήφανοι γιατί είναι και πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας και Βρετανοί και θέλουν να παραμείνουν και ίσως κάποιοι εδώ στο Κοινοβούλιο το ξεχνάνε καμιά φορά και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ε, να βρουν τον τρόπο να διασφαλίσουν αυτό το μηχανισμό ασφαλείας. Το ψήφισμα Φερχόφστατ δεν νομίζω ότι συνεισφέρει τίποτα χρήσιμο στο παρόν στάδιο. Θα θέλαμε να έχουμε μια συντονιστική ομάδα για το Brexit που να είναι πραγματικά δημοκρατική, πλήρως αντιπροσωπευτική και πραγματική πηγή σοφίας και ιδεών και όχι να επαναλαμβάνει μάντρας ε, τα οποία μας έχουν κουράσει να τα ακούμε. Η τελική συμφωνία χρειάζεται τη συμφωνία όχι μόνο του Βρετανικού Κοινοβουλίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, προ όλου ε, εσά που εκπροσωπείτε τι πολιτικέ ομάδε, θέλω να πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τι ε, εντατικέ προσπάθειες. Ε, πρέπει να καταλήξετε σε μία συμφωνία και θα πρέπει πριν από τη συνάντηση του Συμβουλίου στι 18 Οκτωβρίου να έχουν ληφθεί αυτέ οι αποφάσει. Α μην χάσουμε την ευκαιρία να έχουμε μία πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου για όλους τους πολίτες μα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Σιρντεβάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όταν ήμουν καινούριο στο Κοινοβούλιο και άκουσα για το Brexit, άκουσα να μου λένε ε, ότι πρόκειται για την καταστροφή μιας αυτοκρατορίας. το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στη χειρότερη κρίση του εδώ και δεκαετίες. Μια κρίση που θέτει σε κίνδυνο αυτούς που αγωνίζονται για το καθημερινό τους μεροκάματο και όλους τους εργαζομένους. Αυτή η πολιτική δεν είναι προς όφελος ούτε των Βρετανών ούτε των υπολείπων Ευρωπαίων και η κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον το γνωρίζει πολύ καλά. Αυτή η επιχείρηση Yellow Hammer θυμίζει τίτλο ταινίας του James Bond. Η Βρετανική κυβέρνηση ε, αναγνωρίζει με τα έγγραφα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν στο Yellowhammer ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με έλλειψη φαρμάκων αλλά η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή τη στρατηγική που είναι πραγματικά παράνοια μιλάμε για Brexit με ή χωρίς ε, συμφωνία. Ένας νοσηλευτής στη Γερμανία ή στην Πολωνία δεν μπορεί να ξέρει εάν θα μπορεί ε, ε, να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιος που περιμένει να πάρει σύνταξη δεν ξέρει αν θα μπορέσει να πάρει σύνταξη σε περίπτωση που ζει στο, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρει μια οικογένεια στο Μπέλφαστ αν θα μπορέσει να στείλει τα παιδιά της ε, στο σχολείο ή αν πρέπει να φοβάται μήπως συμβεί κάτι στο δρόμο όπως προηγούμενες δεκαετίες γίνονταν ταραχές στους δρόμους. Αν συνεχιστεί αυτή αυτή η πολιτική και αν μιλάμε για ένα σκληρό Brexit, διατρέχουμε τέτοιους κινδύνους. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει η Βρετανική πολιτική να δείξει ότι έχει τη βούληση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Όταν σκέφτομαι την Μεγάλη Βρετανία, σκέφτομαι αυτό που έρχεται στο νου μου από τη λέξη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, με πλούσια ιστορία απικιών, με δημοκρατικά δικαιώματα, με τον John Maynard Keynes, σοσιαλιστές, τον Καρλ Μάξ τον Λονδίνο σκέφτομαι. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Φερχόφσταντ, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για κομικές μορφές τύπου Χάλκ για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εμείς ως αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουμε το ψήφισμα γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπεραμεινθούμε των αξιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίντσης για τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει για να παρεμποδίσουν ε, τους ε, Βρετανούς από το να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα το να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα τρεις-τέσσερις φορές μέχρι να αλλάξει το αποτέλεσμα, το βρίσκεται λογικό. Νομίζω ότι αυτό ε, είναι μια ε, διαστροφή ε, της ε, δημοκρατίας και του δημοκρατικού αποτελέσματος και ένας πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πει πως οι συμφωνίες και λέξεις κάτι θα πρέπει να σημαίνουν. Διαφορετικά ε, δεν υπάρχει νόημα. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πρέπει κάτι να σημαίνει. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Το δημοψήφισμα μίλησε ε, και εδώ αριστερά μου έχω 21 υποστηρικτές του Brexit που είναι το ισχυρότερο κόμμα ε, του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει αυτό. Εκφράζουν τη βούληση του Βρετανικού λαού. Επίσης, αν προσπαθήσουμε να διαβάσουμε το μέλλον. Πριν από μερικές εβδομάδες η κυρία Φόντερ Λάγεν μίλησε για μια κοινή ε, εξωτερική πολιτική ε, ως μια έννοια η οποία θα εισαχθεί και πιστεύω πως είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι πολύ επικίνδυνο δεν μπορεί η Κροατία, για παράδειγμα, να ε, ε, παίρνει εντολέ από την κυρία Φόντερ Λάιν για το τι πιστεύει για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, για τη Μάλτα, για τη ΣΥΠΑ. Αυτό θα χειροτερεύσει τι σχέσει μα στο μέλλον. Φτάνει πια με την προσπάθεια ομοσπονδιοποίηση. Είναι επικίνδυνη αυτή η τακτική. Ο ευρωφουνταμενταλισμός είναι επικίνδυνος. Και όταν να πιστεύει κανείς πως η μόνη λύση είναι να ακολουθηθεί η προσέγγιση Μέρκελ, επίση είναι επικίνδυνη τακτική. Νομίζω ότι χρειάζεται περιθώριο και για άλλες πολιτικές επιλογές και αν δεν το επιτρέψουμε το Brexit θα είναι η αρχή και όχι το τέλος. Χρειαζόμαστε ένα πιο ταχύ τρόπο για αποχώρηση ε, για τις χώρες των οποίων οι λαοί αποφασίζουν πως θέλουν να αποχωρήσουν. Δύο λεπτά η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Ψηφίζουμε σήμερα και κάνουμε τη συζήτηση για το Brexit τη στιγμή που έχουν διακοπεί η λειτουργία του Βρετανικού Κοινοβουλίου της Κάτω Βουλής. Είμαι πεπισμένος ότι οι περισσότεροι από μας λυπούμεθα για το Brexit και εξακολουθούμε εμείς να πιστεύουμε σε ένα Brexit με τάξη. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να συνεσφερούμε στην προσπάθεια βοηθώντας τον Μισελ Μπαρνιέ έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να παρέχει την νομική ασφάλεια και σταθερότητα σε όλους τους πολίτες, τις μικρές επιχειρήσεις, ε, γιατί αυτές οι δύο κατηγορίες μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Η συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει διευκολύνει ε, την αποχώρηση, ε, μια κατανόητη αποχώρηση μια σύγχρονης χώρας ε, και αυτή η ρήξη των δεσμών που δημιουργήθηκαν για 45 χρόνια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία ήταν επίσης ένα σωστό πολιτικό θεμέλιο για την οικοδόμηση των μελλοντικών σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στο μέλλον και μέσω του backstop που είναι ένα σημείο εγγύησης θα έλεγα, ένα δίκτυο εγγύησης ε, πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Λυπάμαι που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει προτείνει νομικά δεσμευτικές και αποδοτικές προτάσεις. Εμείς ε, με υπομονή θα περιμένουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει δυνατότητα κατάληξη σε συμφωνία και θα πρέπει να είναι σαφές ότι η αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα είναι απόλυτη ευθύνη της Βρετανικής κυβέρνησης. Ακόμα και η καλύτερη μορφή προετοιμασίας για την άτακτη αποχώρηση δεν θα είναι παραδιορθωτικά και θεραπευτικά εκ των υστέρων μέτρα. Δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις ούτε για τους πολίτες και τα δικαιώματά τους, ούτε για τα σύνορα στην Ιρλανδία. Και νομίζω ότι ακριβώς μέσω της ε, ε, συντακτικής σύγκλησης των δύο πλευρών πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να καταλήξουμε στην ε, συμφωνία. Κοιτάξτε, καθυστερούμε. Έχουμε 14 επίσης ζητήσει το λόγο μέσα από τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΕ. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να προσπαθήσετε να μην καθυστερείτε ε, και να κάνετε ησυχία. Σίλβα Φερέιρα, ε, ως αντιπρόεδρος θα σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Συζητάμε το Brexit με δημοκρατικό τρόπο, με ελεύθερο τρόπο, με δεκτικό τρόπο, όπως και κάθε κοινοβούλιο θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο πλήρες ε, ε, κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους Βετανούς πολίτες σήμερα. Το κοινό ψήφισμα που κατέθεσαν οι σοσιαλιστές μαζί και με άλλες πολιτικές ομάδες δείχνει το πόσο ενωμένοι είμαστε καθορίζοντας τις θέσεις μας πάνω σε αυτήν την λυπηρή διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Σεβόμεθα πλήρως την βούληση του Βρετανικού λαού. Αν γίνει όμως το Brexit θα πρέπει να γίνει με τακτικό τρόπο, με συντεταγμένο τρόπο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για συντεταγμένη αποχώρηση τα πράγματα θα χειροτερεύσουν ακούσουμε τον κύριο Τζόνσον να λέγει ότι θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ένωση χωρίς ε, το λεγόμενο Ιρλανδικό Δίκτυο Ασφαλείας και ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του Οκτωβρίου παρά τη απουσία συμφωνίας. Αν είναι όμως σοβαρός σε αυτά που είπε ότι θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία τις επόμενες μέρες, θα είχατε τουλάχιστον καταθέσει κάποιες γραπτές προτάσεις ε, εφικτών ρυθμίσεων, νομικά συμβατών. Δεν το κάνατε αυτό και γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι είστε σοβαροί στην προσπάθεια που λέτε ότι κάνετε για να αποφύγετε την άτακτη αποχώρηση. Λοιπόν, αν αποχωρήσετε χωρίς συμφωνία, αυτό θα είναι η απόλυτη ευθύνη στην Βρετανική κυβέρνηση. Και η Κατοβουλή και η Ανοβουλή ενέκριναν ένα νόμο που υποχρεώνει το την κυβέρνηση να ζητήσει παράταση του άρθρου 50 αν δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Δεν δόθηκε καμία εντολή για μη συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία εντολή λοιπόν για μη συμφωνία και από το ε, Βρετανικό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι το ψήφισμά μας διευκρινίζει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την παράταση ε, του άρθρου 50 για να αποφύγουμε το σενάριο της μη συμφωνίας. Ο τρόπος που βλέπουμε την διεύρυνση αυτή ε, θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να βρει λύσεις στα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε έτσι ώστε να ανακτήσει ο Βρετανικός λαός το δικαιώματά του. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκίψον για ένα λεπτό. Σήμερα κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε σοβαρά. Κινδυνεύουμε και εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κίνδυνος είναι να κουραστούμε από την τεράστια αποτυχία που είναι το Brexit και να πιέσουμε να προχωρήσουμε απλώς για να κλείσει το θέμα. Κίνδυνο στη δημοκρατία, στη σταθερότητα, στο κράτος δικαίου, στην ε, κυριαρχία του Κοινοβουλίου οπουδήποτε. Κίνδυνος για τα δικαιώματα των πολιτών. Παροτρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτό το ψήφισμα, να ξεπεράσει την εξάντληση από το Brexit, να, επεκτεί, να δώσει δυνατότητα επέκταση προθεσμίας στο άρθρο 50 για να έχει το χρόνο ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να ε, καταφέρει να ξεπεράσει τα όσα έκανε ο δικτάτορας αυτός, ο οποίος ε, στέρισε τη φωνή από το μεγάλο δημοκρατικό θεσμό που είναι το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το Brexit σας είναι καταστροφή και αξίζει να πάρετε όσο χρόνο χρειάζεται για να το σταματήσετε. Για δύο λεπτά ο κύριος Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, καλημέρα. Το Brexit ε, μας έχει εκνευρίσει από την αρχή και αυτό είναι λυπηρό. Και να σας πω πως από την πλευρά της Σκοτίας το θεωρούμε και φοβερά άδικο. Εμείς ψηφίσαμε να μείνουμε στην οικογένεια των ε, εθνών μας. Το ίδιο έκανε και η Ιρλανδία. Η ειρηνευτική διαδικασία εκεί είναι ιερή και θα πρέπει να προστατευθεί. Το... Οι Σκοτσέζοι δεν έχουν μαζί σας κανένα πρόβλημα. Μόνο το Westminster το οποίο δεν αξίζει ε, να έχει το ρόλο που έχει σε ένα σύγχρονο και προοδευτικό κόσμο. Δεν θέλω να σας κουράσω με τα εσωτερικά μας προβλήματα. Εσείς λυπάμαι που το λέω αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τους ομιλητές που σας έστειλαν. Και προσπαθώ σήμερα να πω το εξή. Ας αποφύγουμε ένα τεράστιο σφάλμα όλοι μας σήμερα. Ακούω το επιχείρημα κάθε χρόνο που μας λένε στη χώρα μου ναι να παραδώσουμε τον Brexit, να γίνει το Brexit, να ξεπεράσουμε το Brexit, να το αφήσουμε πίσω μας το Brexit και ακούω και εσά να έχετε πια βαρεθεί τις βρετανικέ ανοησίε. αν σας βοηθά αυτό και εγώ έχω βαρεθεί. Και καταλαβαίνω πως θέλετε μια συντεταγμένη διαδικασία για να ελαφρύνετε τα προβλήματα που θα φέρει το Brexit. Λυπάμαι συνάδελφοι, οι ειδήσει που φέρνω είναι απογοητευτικέ. Δεν υπάρχει καλό Brexit, δεν υπάρχει βιώσιμη λύση οι άνθρωποι με τους οποίους έχετε να κάνετε που είναι ε, τα άδεια ανδρίκελα του συντηρητικού κόμματος λείπουν από την αίθουσα αυτή και οι αντικαταστάτες τους δεν θέλουν μια Ευρώπη που να λειτουργεί. Και αν κάνουν Brexit θα το κάνουν για να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια τακτική καταστροφής της γης ε, στη χώρα μας και θα υποφέρουν οι Ουαλοί, οι, οι Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί. Θα κάνουν απίστευτο dumping. Δεν υπάρχει καλό Brexit. Δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να στηρίξω το ψήφισμα παρόλο τις καλύτερες προσπάθειες και την καλή πίστη που έχετε δείξει γιατί δεν πιστεύω που η συμφωνία αποχώρησης θα φέρει ε, κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αντιστρέψουμε ως κοτσέζι το Brexit. Σας παρακαλώ πολύ το χρόνο αυτό να μας τον δώσετε. Are you finished? Τελειώσατε να φωνασκείτε. Η πρόεδρος ρωτάει ποιος κάνει αυτά τα σχόλια εκτός μικροφώνου. Εγώ έχω τον έλεγχο, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπέκ, τρία λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, η Μεγάλη Βρετανία μπροστά στο χάος έτσι κινδυνολογούν ε, τα μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία, όπως και η ιστερία πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. Ε, Παρ' όλα αυτά, όντως υπάρχουν σοβαρές συνέπειες που απειλούν ε, το μέλλον μας. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η τρίτη σε μέγεθος εξαγωγική αγορά για τη Γερμανία και μαζί με τις ΗΠΑ η πιο κερδοφόρος. Για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά. Σε περίπτωση σκληρού Brexit κινδυνεύουν να χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επιπλέον υπάρχει και το κόστος από την απώλεια της καθαρής συνεισφοράς της Βρετανίας 10 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ και η Γερμανία που πάντα σέβεται τους νόμους θα πληγεί περισσότερο. Οπότε γιατί αρνείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα φιλικό διαζύγιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύτηκε καλή την πίστη, ίσω υπερβολικά καλή την πίστη, ε, όταν συμφώνησε με όλα τα αιτήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για τα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το νόμο περί διαζυγίου, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε ε, δημιουργώντας αυτό το θέμα του Ιρλανδικού backstop. Αλλά σοβαρά τώρα, ποιος πιστεύει ότι κάποιοι σποραδικοί ή ηλεκτρονικοί τελωνιακοί έλεγχοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν ε, στην ε, αναβίωση ε, της βίαιης τρομοκρατίας στην Ιρλανδία ούτε καν ο Μισελ Μπαχνιέ που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το backstop για να κρατήσει τη Βρετανία σε μια διαρκή τελωνιακή ένωση ή να την υποχρεώσει σε ένα δημοψήφισμα. Εναντίον όλου του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου και εναντίον ε, κάθε πολιτικά ορθής ε, άποψης που επικρατούσε στο παρελθόν, ο λαός της Βρετανίας ε, ψήφισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πλειοψηφία 52 προς 48%. Ίδια πλειοψηφία δηλαδή με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη θέση της ε, εκλεγής σας ε, Πρόεδρου της Επιτροπής, κυρίας Φόντερ Λάιεν. 17,4 εκατομμύρια Βρετανοί πολίτες ψήφισαν υπέρ του Brexit, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός Βρετανών πολιτών που ψήφισαν, που πήγαν ποτέ να ψηφίσουν για οτιδήποτε. Ο Μισελ Μπαχνιέ είναι έξυπνος ε, και επιδέξιος διαπραγματευτής, αλλά προσπαθεί να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο υποτελές κράτος ή εναλλακτικά να διακινδυνεύσει τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά και τα δύο αποτελέσματα είναι απαράδεκτα. Ένα λεπτό, κύριος Λούντγκριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τον Brexit υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένου Βασιλείου και οι δύο πλευρές ε, δυσκολεύονται να καταθέσουν χρήσιμες προτάσεις. Πριν από κάποιε δεκαετίε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήθελε να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγου παρόμοιου όπω και τώρα στο Brexit. δεν ήθελε τελωνιακή ένωση. Και θα προτιμούσε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, επιδιώκοντας το δίκαιο ανταγωνισμό. Θα ήταν προτιμότερο να έχει μια συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μαζί με τη Σουηδία. Τώρα οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν και θα πρέπει να αποδεχθούμε αυτό που ψήφισαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με το χρόνο, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Άντερσον, 1,5 λεπτό. Το Ιρλανδικό διαβατήριο μου λέει ότι έχω τα δικαιώματα σαν κάτοικος του νησιού της Ιρλανδίας να ανήκω στον Ιρλανδικό έθνος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι Ιρλανδοί στη Βόρεια Ιρλανδία, αν θέλουμε μπορούμε να είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το backstop έχει σαν στόχο να προστατεύσει το σύνολο της ε, οικονομίας στο νησί, να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών και να μας προστατεύσει από την επιβολή μέτρων που εμείς δεν θέλουμε. Είναι σημαντικό το κοινοβούλιο αυτό να αναγνωρίσει όπως λέγεται στο ψήφισμα την ελεύθερη επιλογή, τον σεβασμό της ελεύθερης επιλογής της πλειοψηφίας του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας και του δικαιώματός του σε αυτοδιάθεση όπως το λέει και η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και όπως το προβλέπει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι η λύση στο πρόβλημα του Brexit είναι η επανένωση της Ιρλανδίας. Και νομίζω ότι η λογική λέει ότι υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ της επανένωσης και η συμφωνία ακριβώς της Μεγάλης Παρασκευής δίνει την δυνατότητα επιστροφής στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας ο κύριος Φαράζ. Ακούσαμε διάφορα από τον κύριο Μπαρνιέ και τον κύριο Γιούνκερ που είπαν ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία για το backstop πριν από το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό το παρουσιάζουν σαν μια διαπραγματευτική νίκη, αλλά να πω ότι η συμφωνία αυτή και η συνθήκη αυτή είναι θα έλεγα ακόμα και αν υπάρξει ή δεν υπάρξει backstop είναι μια κακή λύση εξακολουθούμε να ελέγχουμε τα πάντα και στην ουσία η Μεγάλη Βρετανία θα είναι σε μειονεκτική θέση και δεν θα υπάρχει καλή πίστη ανάμεσά μας στο μέλλον. Ε, αφεθήκαμε ε, στο έλεος σας ουσιαστικά εμείς στην Βρετανία και το μήνυμα που στέλνουμε πια είναι ότι να μην μας λέτε ότι υπάρχει καλή πίστη γιατί ε, παραπέμπεται τότε στα αστεία τα οποία είπε ο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου που προσπάθησε να μειώσει τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και ο πρόεδρος Μακρόν στο Παρίσι. Το να παραμένουμε παγιδευμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο στόχος του Μπαρνιέ, το είπατε κύριε Μπαρνιέ και σήμερα το πρωί. Θέλετε να παραμείνουμε έγκλειστοι στην τελωνιακή ένωση. Εμείς θέλουμε να φύγουμε όμως, θέλουμε να φύγουμε από την αγορά σας. Θέλουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, θέλουμε να γίνουμε πιο πλούσιοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ανήκουμε στην ευρωπαϊκή σας αυτοκρατορία κύριε Φερχόφστατ. Εμείς θέλουμε ένα ξεκάθαρο Brexit χωρίς όρους και όταν το πετύχουμε αυτό και όταν το κάνουμε αυτό θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ο κύριος Γκοντζάλης Πόνς για 1,5 λεπτό. Όταν ήμουν ε, φοιτητή, νέος, και άρχισα να ανακατεύουμε την πολιτική, θεωρούσα ύψιστο υπόδειγμα του τι είναι η δημοκρατία, του Ηνωμένου Βασίλειου. Αυτό δεν συμβαίνει πια. Είναι μια σκιά του εαυτού του το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί υπάρχουν πολιτικοί όπως ο Νάτζελ Φάραντζ. Σήμερα από το Ηνωμένο Βασίλειο περνά τι πιο σκοτεινές ώρες από τον καιρό του πολέμου, κλείσαν τη Βουλή. Τις τελευταίες στιγμές της διαπραγμάτευσης το δικό μας κοινοβούλιο είναι ανοιχτό, το Βρετανικό, το έχουν κλείσει. Και γι' αυτό σήμερα όλοι εδώ πρέπει να μιλάμε αγγλικά, γιατί εκπροσωπούμε όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά και το βρετανικό λαό. Σήμερα εδώ είναι ο βρετανικός οίκος της δημοκρατίας. Σήμερα έχουν πάρει τα ενία στο Ηνωμένο Βασίλειο λαϊκιστές πολιτικοί οι οποίοι έχουν τα δικά τους όρια και οι οποίοι προσπαθούν ε, να κάνουν μια διαπραγμάτευση και εμείς από την πλευρά μας έχουμε διαπραγματευτεί όσο πιο καλά μπορούμε. Με καλή βούληση. Είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτέ και ο κύριο Μπαρνιά και ο κύριο Γιούμκερ, αλλά είναι και έντιμοι πολιτικοί. Μπορούν να πούν τα ίδια οι Βρετανοί πολιτικοί. Εμεί να του δώσουμε μια επέκταση προθεσμία, αλλά θα πρέπει να μα εξηγήσουν το γιατί και το μέχρι πότε. Δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας. Παροτρύνω τον Πρωθυπουργό να σεβαστεί το Βρετανικό Κοινοβούλιο και τον παροτρύνω να σεβαστεί και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Γιατί το Brexit δεν είναι μόνο καταστροφή. Είναι και το πιο επίκαιρο θέμα αυτή την εποχή. Ο κύριος Κόρμπετ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, είναι χαόδη και χαοτική η πολιτική κατάσταση Βρετανία αυτή τη στιγμή. Αλλά οι συνάδελφοι δεν θα πρέπει για οποιαδήποτε στιγμή να πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργό αυτό και εκείνοι εκεί που κάθονται εκεί εκπροσωπούν ολόκληρο το Βρετανικό λαό. Όχι, και δεν θα πρέπει να επιτρέψουν ε, στον ε, κύριο Τζόνσον να δηλώνει πως ζητά ε, συμφωνία, μα δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση στο τραπέζι και οι ιδέες που παρουσιάζει κατά καιρού είναι ιδέες τις οποίες δεν μπορούν να γίνουν δεκτές ούτε εδώ ούτε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά κατευθύνεται προς ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Αλλά το Βρετανικό Κοινοβούλιο νομοθέτησε για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Απαιτεί από αυτό να ζητήσει επέκταση της προθεσμίας και να μην επιτρέψει το Brexit χωρίς συμφωνία. Και η πλειοψηφία στη Βρετανική Βουλή αυτή τη στιγμή, και θυμηθείτε το γιατί αυτή τη στιγμή έχει χάσει υπουργού, έχει διώξει μέλη, είναι μια κυβέρνηση μειοψηφία. Και κάθε ένα κόμμα στην αντιπολίτευση. Η εργατικοί, οι φιλελεύθεροι, οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί θέλουν καινούριο δημοψήφισμα. Και νομίζω ότι αν γίνει δημοψήφισμα για το no deal που προτείνει ο κύριος Τζόνσον, ε, θα κάναμε εκστρατεία υπέρ της παραμονής. Οπότε όσο και να εκνευρίζεστε από τη Βρετανική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σας, θυμηθείτε το αυτό. Δεν είναι οι Βρετανοί πολίτες. Έχει αλλάξει και μετακινηθεί η κοινή γνώμη. Χρειάζεται νέο δημοψήφισμα, δικαιολογείται γιατί γιατί το Brexit που παρουσιάζουν δεν έχει καμία σχέση με τα όσα μας παρουσίαζαν εκείνοι εκεί όταν κάναμε την εκστρατεία. Μας έλεγαν ότι θα είναι εύκολο, πως θα εξοικονομήσουμε χρήματα που θα πάει στο ΕΣΥ. Κοστίζει μια περιουσία. Μας είπαν πως θα είναι καλό για τη Βρετανική οικονομία. Και το αντίθετο ισχύει. Γι' αυτό όσοι έχουν ψηφίσει να αποχωρήσουν έχουν δικαίωμα να πούν δεν είναι αυτό που μου υποσχεθήκατε, δεν είναι για τούτο που ψήφισα. Έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε και είναι σωστό να δώσουμε στο Βρετανικό λαό το δικαίωμα να ξαναποφασίσει. Και σας παρακαλώ δώστε μας αυτή την επέκταση, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, έχει λήξει ο χρόνος σας. Για ένα λεπτό η κυρία Λόγκ. Κύριε Πρόεδρε, εξελέγει ω πολιτικό ε, όλων των κοινοτήτων για του πολίτε τη ε, Βορείου Ιρλανδίας και μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ του να παραμείνουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι σημαντικό το να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κομμάτι της κοινή μα ταυτότητα, ενώνει όλου τους πολίτε, και τους ενωτικού και του μη ενωτικού. Η Συμφωνία της μεγάλη παρασκευή βασίζεται σε συνεργασία και πρέπει να προστατευθεί η κυβέρνηση ε, από πλευρά του DUP αρνήθηκε να μα ακούσει. Όταν ήταν αντίθετη με τη συμφωνία τη μεγάλη παρασκευή το 1988 δεν συμφωνούσε με την γνώμη των πολιτών και δεν άκουσε τη γνώμη των πολιτών όπω και τώρα δεν ακούει τη γνώμη των πολιτών. Ένα Brexit χωρί συμφωνία θα είναι καταστροφικό για τη Βόρεια Ιρλανδία. Μην ακούτε αυτού που λένε ότι χωρί συμφωνία δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ε, ακούστε αυτού που δουλεύουν και από τι δύο πλευρέ των συνόρων που ξέρουν τι συμβαίνει επί τόπου. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθεί να αποφύγει, πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει μια συμφωνία, μια έξοδο χωρίς συμφωνία. Εκτιμούμε την υπομονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε τον Brexit, όχι μόνο να γίνει, αλλά να γίνει σωστά. Could I just... Θέλω να ρωτήσω τουλάχιστον αυτή την, να ζητήσω από αυτή την πλευρά της αίθουσα, αν μιλάτε μεταξύ σας τουλάχιστον χαμηλόφωνα γιατί ενοχλείτε όλη την αίθουσα. Τώρα για δύο λεπτά η κυρία Σκοτ Κέιτ έχει το λόγο. Το θέμα του Brexit είναι θέμα ελέγχου. Ο Τζόνσον και οι ακολουθοί του δυστυχώς έχασαν τον έλεγχο της χώρας τους διέκοψαν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, μια παράλογη κατάχρηση εξουσίας ε, που είχε να συμβεί από τον 18ο αιώνα και είδαμε και τη συμπεριφορά του Τζόνσον στο Λουξεμβούργο πρόσφατα. Λοιπόν, στην ουσία παίρνουν τον έλεγχο από τους κοινοβουλευτικούς, παίρνουν τον έλεγχο από αυτούς που στηρίζουν το δίκαιο, ε, το Brexit δεν ενισχύει τον λαό, δεν ενισχύει την κυβέρνηση, ενισχύει τους πλούσιους ε, μια μικρή κατηγορία πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για εδώ ακριβώς ε, τίθενται τα θέματα προστασίας του καταναλωτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εμείς ένα αγώνα προς τα κάτω. Ε, δεν θα επιτρέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει ο βρώμικος Ευρωπαίος. Δυστυχώς ε, ε, και οι εκπρόσωποι, οι πολίτες μάλλον των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει και αυτοί αντικείμενο εκβιασμού από πλευράς της Βρετανικής κυβέρνησης. Πρέπει να ληφθούν θετικά μέτρα για την προστασία της δημοκρατίας. Λέει το ψήφισμά μας ότι περιμένουμε εμείς από το, Ηνωμένο από το Συμβούλιο να δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο την, παρά... την παράταση την οποία επιθυμεί. Μόνο εμείς μπορούμε να αντισταθούμε στην τυραννία του Τζόνσον και αυτών που τον ακολουθούν. Ε, χρειαζόμαστε χρόνο για να πάρουμε πίσω την εξουσία από τους υπερπλούσιους και τους ολιγάρχες. Τότε μόνο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη του Brexit. Ευχαριστώ. Με το δημοψήφισμα, μια ιστορική ημέρα, 51,8% επέλεξαν να φύγουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε μέρα από τότε η πολιτική ελίτ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κρατούν ομήρους τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Ιρλανδίας. Είναι δεσμευτική η συμφωνία του, η απόφαση του δημοψηφίσματος ε, και πρέπει να τηρηθεί. Μπορεί κάποιοι πολιτικοί να πιστεύουν ότι αν εμποδίσουν το Brexit ε, θα πράξουν σοφά, αλλά δεν μπορούν να το επιβάλλουν σε αυτούς που έχουν ε, τη δύναμη. Μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κηρύσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε τρίτες χώρες αλλά οι δημοκρατικές αρχές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται μόνο όταν αντιστοιχούν στην ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η δυνατότητα του να είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε συνοδεύεται από δυνατότητα να αποχωρήσει. Αλλά οι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει. Και ο κύριος Φερχόφστεντ και οι συνάδελφοί του προσπαθούν να κρατήσουν όμοιρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει πει ότι μπορεί να επιτύχει το Brexit, αλλά η Βουλή των Κοινοτήτων συνεχώς τον υπονομεύει και μάλιστα πρόσφατα ψήφισε ένα νόμο να κηρύξει παράνομο το Brexit χωρίς συμφωνία. Θα μπορούσε ο Τζόνσον να διαπραγματευτεί μια διαφορετική συμφωνία ή να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία. Δεν θα κρατήσετε ομήρους ε, τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αγνοώντας το ποιος ε, ε, ευθύνεται ε, για αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούσει τους λαούς και να τηρήσει την κυριαρχία των λαών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ζαραντήλ. Ευχαριστώ πολύ. Έξι εβδομάδες μέχρι το Brexit και αν δεν συμβεί τίποτα, 31 Οκτωβρίου αποχωρεί το Ενωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κόσμος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σφάλουν, γιατί πιστεύουν πως υπάρχει συμφωνία και ότι μόνο κάποιοι ταραξίες από το Ηνωμένο Βασίλειο φρενάρουν αυτή τη συμφωνία και θα πρέπει να λογικευθούν. Αυτό δεν ισχύει, δεν αληθεύει, δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε μόνο ένα σχέδιο, το οποίο τρεις φορές έχει καταψηφιστεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων και που η τρέχουσα ε, νομιμοποιημένη και νόμιμη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν δέχεται χρειάζονται δυο για να χορέψει κανείς ταγκό. Αλλά νομίζω ότι εμείς εδώ χορεύουμε μόνοι μας. Το πιο λογικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει την εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία αυτή. Αλλιώ, σε έξι εβδομάδε θα φτάσουμε στη μη συμφωνία με καταστροφικέ συνέπειε για τι οικονομίε μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάναγκαν για ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου, ο κύριος Φλάναγκαν. Πρώτον, Καταρχήν να δούμε πώς λειτουργούν τα μικρόφωνα. Πρώτον λοιπόν επανέρχομαι. Θα πρέπει καταρχήν να σεβαστούμε τις θέσεις όλων και να σεβαστούμε το ότι ψήφισε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει. Και αυτοί που θα αποχωρήσουν θα πρέπει να σεβαστούν ότι αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα για όσους ζουν στις περιοχές που συνορεύουν. Αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση είναι το backstop και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Και τότε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα ε, δοκιμαστεί γιατί μέχρι σήμερα έχει μείνει στις λέξεις. Μας λέει κάθε φορά ο Ιούγκερ πως χρειαζόμαστε αλληλεγγύα. Οι εξαγωγές ε, της Ιρλανδίας είναι μισό εκατομμύριο ε, τόνοι βοηίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να βρούμε άλλες αγορές. Να πάνε λοιπόν στους Ευρωπαίους γείτονε. Έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, αν το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει χωρίς συμφωνία, τότε η Ιρλανδία χρειάζεται μια νέα αγορά. Εμείς 300.000 είχαμε εισαγωγέ βοή από τι χώρε του Μερκοσούρ πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρχουμε συμφωνία, ο νέο επίτροπο ε, ο Φιλ Χόγκαν για το εμπόριο να κλείσει την κάνουλα για αυτές τις εισαγωγές βοή από το Μερκοσούρ αν πραγματικά εννοούμε τις λέξεις που λέμε για την αλληλεγγύη. Κυρία Ντότς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω πως ε, μια συντεταγμένη αποχώρηση είναι η καλύτερη και προτιμόμενη λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ενωμένο Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα για τους γειτονές μας στην δημοκρατία της Ιρλανδίας. Πιστεύω πως αυτό είναι προς συμφέρον μας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το πετύχουμε. Όμως, η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να βλάπτει τα συνταγματικά και οικονομικά ε, συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Ιρλανδίου ως τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δημοκρατικό καθήκον αυτό και το backstop διακυβεύει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επιβεβαιώσει πολλές φορές πώς θα ε, σεβαστούμε τη συμφωνία του Belfast. Και σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Γιούνκερ και ο κύριος Μπαρνιά αναφέρθηκαν σε αυτή τη συμφωνία. Βασική αρχή είναι η ισοτιμία των δύο παραδόσεων και κοινοτήτων στην ε, στα δύο κομμάτια ε, αυτά της Βορείου Ιρλανδίου. Δηλαδή, οι εθνικιστές και οι προτεστάντες θα πρέπει να τύχουν τις ίδιες μεταχείρισης. Ο κύριος Αχέρν, πρώην Πρωθυπουργός που είχε οικοδομήσει αυτή τη συμφωνία. Μίλησε για τη συμφωνία της ισότιμης μεταχείρισης και είχε πει πως οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους ενωτικούς γιατί στη συμφωνία αυτή θα πρέπει να καλύψουμε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Η επιστολή που έχει σταλεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και που δημιουργεί τη δήλωση 5 του ψηφίσματος δεν έχει υπογραφεί ούτε έχει στηριχθεί από οποιοδήποτε μέλος ε, του ε, Βορειοελλανδικού Κοινοβουλίου που να προέρχεται από τους ενωτικούς και στις εκλογές ε, εμείς υποσχεθήκαμε πως θα απορρίψουμε το backstop. Το 81% των ενωτικών είναι κατά του backstop. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικό με το backstop κύριε Μπαρνιέ. Και εσείς δεν μπορείτε να νύπτετε τη σχήρα σας. Ούτε μπορούμε να ε, ε, γεμίσουμε την Βόρεια Ιρλανδία με νομοθεσία την οποία δεν έχει τρόπο να επηρεάσει. Πρέπει να είμαι πολύ αυστηρή, κυρία Ντότς. Με συγχωρείτε, σας παίρνω το λόγο, κύριο Ταγιάννη, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, της οποίας είμαι πρόεδρος, έδωσε την δυνατότητα στις οργανώσεις των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Ιρλανδών ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, ακούσαμε επίσης και τα αιτήματα των Βρετανών υπηκών που ζουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει φωνή σε αυτούς που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες και συμπατριώτες μου που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ είμαστε ο χώρος της δημοκρατίας. Εδώ είμαστε ο χώρος που θα υπερασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών έτσι ώστε να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τους λαούς της Ευρώπης. Εμείς ζητήσαμε να πάμε και στα σύνορα ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα τι θα πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ειρήνη είναι σημαντικό το backstop. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε και από τις μυστικές υπηρεσίες των Βρετανικών, τις Βρετανικές είναι ανησυχητικέ. Ε, πρέπει να προστατεύσουμε μέσω ενός ευέλικτου τύπου συνόρων τη γεωργία μας, τις επιχειρήσεις. Θυμηθείτε τι έγινε με τις τρελές αγελάδες. Ε, χωρίς ε, ε, μια σωστή ρύθμιση η Ευρώπη θα διατρέξει πάρα πολλούς κινδύνους και γι' αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας. Ο κύριος Μποναφέ ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φτάνουμε στις 31 Οκτωβρίου και ο κύριος Τζόνσον δεν έχει κάνει καμία πολιτική πρόταση η οποία να μπορέσει να συζητηθεί σοβαρά. Αυξάνεται λοιπόν η πιθανότητα άτακτης αποχώρησης την οποία φαίνεται να, προτιμά και η ηγεσία του συντηρητικού κόμματος και κάποιες πρωτοβουλίες του Κόρμπιν για να απαγορεύσει αυτήν την καταστροφική διέξοδο ε, έχουν βοηθήσει. Εμείς και το κόμμα μας, το Δημοκρατικό Κόμμα, θέλουν να βοηθήσουν ε, τρία εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων 700.000 Ιταλοί και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν το ζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά και θα εγκρίνουμε την παράταση αλλά μόνο για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άτακτη αποχώρηση. Ευχαριστώ κύριο Σκέλχαν. Θέλω να υποστηρίξω το ψήφισμα, δέχομαι εγώ την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποχώρηση, αλλά υπάρχει μια υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποδεχθεί το τι προβλέπει η δημοκρατική διαδικασία που αποφασίστηκε στη Βόρεια Ιρλανδία από το 1998 και μετά από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η Συμφωνία προβλέπει για την, τον αμοιβαίο σεβασμό, προβλέπει την αμοιβαία εκτίμηση και προβλέπει και ειδικότερα μέτρα στον τομέα της οικονομίας. Ένα σκληρό Brexit θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ελευθερίες των πολιτών και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο αθλητικό ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από το Ηνωμένο Βασίλειο να παραδεχθεί ότι έχει την νομική υποχρέωση να διαφυλάξει την ακαιρεότητα της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής μιας κατεξοχήν ειρηνευτικής συμφωνίας. Δέχομαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να φύγει, αλλά δέχομαι και το, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Η κυρία Εύανς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι εδώ 20 χρόνια. Ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη πρόκληση. Τώρα όμως αντιμετωπίζουμε τους πιο δύσκολους καιρούς. Το Westminster απέτυχε και δεν βοηθά την Ουαλία, δεν βοηθάει το λαό. Είναι κοινοβούλιο στο όνομα και θα ήθελα να δείτε και ότι άλλο συμβαίνει. Τους τελευταίους μήνες εγώ έχω κάνει πορείες με χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ουαλία στηρίζοντας την ανεξαρτησία. Και αυτή η στήριξη όλο και αυξάνεται το 40% των Ουαλών λέει πως θα στήριζε την ανεξαρτησία της Ουαλίας εάν μπορούσε με τον τρόπο αυτό η Ουαλία να παραμείνει στο, στην Ενωμένη Ευρώπη. Θέλουμε εμείς να χαράξουμε το δικό μας μέλλον και για να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή θα πρέπει να ξαναστραφούμε στο λαό μέσω ψηφίσματος και χρειαζόμαστε χρόνο. Εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση και για το μέλλον της Ουαλίας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βιλίμσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα θέλω να εκφράσω το ότι δεν καταλαβαίνω ότι δύο μεγάλοι διαπραγματευτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διακηρύσουν ότι επηρεάζουν την κοινή γνώμη και δεν είναι σε θέση να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Υπάρχουν δύο μεγάλα στρατόπεδα βλέποντας και αυτή την αίθουσα. Οι μεν λένε ότι το Brexit είναι καλό, οι άλλοι λένε ότι το Brexit είναι κακό. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει σημασία τι λέτε. Σημασία έχει αυτό το οποίο πιστεύω εγώ, αυτό πιστεύει ο λαός της Βρετανίας. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε σεβασμό, να δείξουμε σεβασμό για την πλειοψηφία του βρετανικού πληθυσμού που αποφάσισε επ' αυτού. Και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αυτό θέλουν να κάνουν. Να έχουμε ένα αποτέλεσμα λοιπόν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου που να είναι αποτελεσματικό, επαγγελματικό και όχι αυτό το θέατρο που παίζουμε εδώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Μπουρζουά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν συμμετέσχομαι απευθείας στην Συντονιστική Επιτροπή αλλά η αντιπροσωπεία της Φλάνδρας ε, θα ψηφίσει υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε μια συμφωνία. Και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις προσπάθειες με την απαραίτητη ευελιξία, τηρώντας τις αρχές για το μηχανισμό ασφαλείας, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς. Όσον αφορά τις μελλοντικέ σχέσεις, τόνισε ο κύριος Μπαχνιέ ότι δεν υπάρχει μόνο το εμπόριο, υπάρχει το θέμα της άμυνας, της ασφάλειας, της έρευνας, της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, η γαλάζια οικονομία και πρέπει να τονίσουμε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι Κυρία Ντέλη, το Brexit δεν είναι μόνο για τρελούς Βρετανούς. Το Brexit ε, είναι κάτι που δείχνει την αποτυχία της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Και ηρωνικά αυτό είναι δρεωμένο και στην ε, άρχουσα τάξη στη, Βρετανία. Υπονομεύει ε, τις δημόσιες υπηρεσίες και ας ε, μην ε, κοροϊδευόμαστε. Για τη δημοκρατία μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να τηρεί τις ασχέσεις της δημοκρατίας. Η Βρετανία κανιβαλίζει τη χώρα της και σίγουρα δεν συμφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε σκληρά σύνορα. Πρέπει τα δικαιώματα να τηρηθούν, τα δικαιώματα των λαών που πιστεύουν στην αλληλεγγύη, στην ειρηνική Ευρώπη. Όλοι αυτοί που έχουν αυτά τα πιστεύω όπως και εγώ, θα πρέπει να σταματήσουμε να τηρούμε την πολιτική νεοφιλελευθερισμού. Ευχαριστώ. Κύριος Ντόμπνη. Πολλά μας είπατε σήμερα για τον αυτοκράτορα Φερχόστατ και την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία που θέλει να οικοδομήσει. Είπατε πως ο κύριος Τζόνσον ή η κυρία Doubtfire. Ε, εσείς είσαστε ο Dark Vader της Ευρώπης. Και η εθνική δημοκρατία πεθαίνει στα πόδια σας. Για την αυτοκρατορία να σας πω πως είμαστε 17,4 εκατομμύρια που θα επιτεθούμε πόσα χρόνια πριν πέθαναν οι προγονεί μου στο ευρωπαϊκό έδαφος για να δώσουν τη μάχη κατά του φασισμού. Σήμερα θα απελευθερώσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δις το μήνα πληρώνουμε τα τρία, τελευταία τρία χρόνια για τον τίτλο του μέλους και μας αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση. Ε, άμα θέλετε ίσως κανόνες παιχνιδιού, δεν θα ήθελα καθόλου να παίξω ποδόσφαιρο μαζί σας κύριο Μπαρνιέ. Στημένο θα ήταν το παιχνίδι. Εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύετε στη δημοκρατία. Σήμερα ε, θέλετε να ψηφίσουμε για να πούμε πως είναι λυπηρό γεγονός το Brexit. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Je ne regrette rien. Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mr. Kelly, for Κύριε για 1,5 λεπτό. Ίσως μετά από χρόνια ιστορικοί θα περιγράφουν το Brexit ως το φοβερό μούτρωμα σάλκ του φοβερού χάλκ. Γιατί στις 31 Οκτωβρίου, ό,τι και να γίνει, παρόλες οι επιπτώσεις, θέλει να φύγει. Ό,τι και συνέπειε να έχει αυτό για το νησί τη Ιρλανδίας, για την οικονομία της και για την ειρήνη. Και γι' αυτό είμαστε τόσο ευγνώμονες στην Ιρλανδία για την αλληλεγγύη που δείχνουν. Όσο όμορφα το εξέφρασαν σήμερα το πρωί ο κύριος Γιούνκερ και ο Μπαρνιέ. Είπε ο κύριος Γιούνκερ πως η αλληλεγγύη θα δοθεί στι χώρε που περισσότερο επηρεάζονται και νομίζω ότι αυτό που είπατε ήταν ξεκάθαρο και ο κύριος Μπαρνιέ είπε πως υπάρχει ανάγκη ε, να έχουμε ένα είδος ε, backstop, μια δυνατότητα για δίκτυα ασφαλείας. Υπάρχει και μία ακόμα επίπτωση του άτακτου Brexit μετά από τη συμφωνία του, ε, τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής η σχέσεις μεταξύ μας με το Ηνωμένο Βασίλειο βελτιώθηκαν και ήρθε και η βασίλισσα στο Ντάμπλιν. Ε, αυτά ε, δυστυχώς τώρα έχουν αντικατασταθεί από την υποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνη. Ζητώ να επεκταθεί το άρθρο 50 και αισθάνομαι τη βεβαιότητα μετά από ακούω πως θα επιτραπεί και θα δώσουμε στον κύριο Τζόνσον τη δυνατότητα να παρουσιαστεί με τη μεγάλη γκάμα και πλειάδα δυνατοτήτων που είπε στον Πρωθυπουργό μας πως έχει στο μυαλό του. Και Ελπίζω πως ο κόσμος αφού ψηφίσει θα πάρει την εξουσία από τα χέρια αυτών των ε, ε Brexiteers οι οποίοι ε, αυτή τη στιγμή συνηγορούν υπέρ της μη συμφωνίας Είμαι και Αγγλίδα και Γερμανίδα. Έχω και τις δύο επικότητες και είναι πολύ σημαντικό το θέμα για μένα, λέει η κυρία Μπάρλι. Και βεβαίως συναισθηματικά ε, το δύσκολο για μένα είναι το backstop. Αυτό το οποίο δεν λέμε συχνά είναι πως είναι προσωρινή λύση μέχρι να υπογραφεί η τελική συμφωνία. Οπότε τι σας δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Πρόβλημα είναι γιατί δεν υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη και το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, πολλοί φοβούνται πως θα τους εγκαταλείψουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πάντα και κάποιοι άλλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν την απόλυτη βεβαιότητα πως δεν θα έχουμε σκληρά σύνορα μεταξύ ΙΡΕ και Βορειοϊρλανδίας. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο το θέμα. Και με την Ιρλανδία πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνουμε θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που προτείνουν στην Βρετανία και κάποιοι εδώ πολιτικοί. Δηλαδή, να είμαστε όλο και πιο επιθετικοί, να χρησιμοποιούμε όλο και πιο πολλές ε, εκφράσεις από, ε, που να παραπέμπουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το λέω αυτό γιατί είμαι και Βρετανή και Γερμανίδα. Θα πρέπει να είμαστε καλοί γείτονες και να παραμείνουμε καλοί γείτονες και στο μέλλον. Για ένα λεπτό, κυρία Λουαζό. Να ευχαριστήσω τον Γιούνκερ και τον Βαρνιέ που είναι μαζί μας σήμερα στο κοινοβούλιο το οποίο έχει την δυνατότητα να σας ακούσει ε, και να συζητήσει το Brexit χωρίς κανένας να το απειλεί για διακοπή των εργασιών του. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θίξουμε την νήσο της Ιρλανδίας με ένα τείχος ή με την επιστροφή στη βία. Ε, ποτέ δεν θα θελήσουμε να απειλήσουμε την ακαιρεότητα του Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών της. Ε, το κοινοβούλιο μας πάντα λέει αυτό το οποίο επιθυμεί και η στάση μας απέναντι στο Βρετανικό λαό είναι στάθη σεβασμού. Αγνοούμε όμως το τι επιθυμεί η Βρετανική κυβέρνηση. Αγνοούμε αν θα ζητήσει ε, περαιτέρω παράταση για τον Brexit, αν έχει λόγους να το κάνει. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν λέει ούτε πότε, ούτε πώς, ούτε ε, εν πάση περιπτώσει αν πραγματικά θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τον τρόπο που θα το κάνει. Καλό είναι να πει επιτέλους την αλήθεια η Βρετανική πλευρά. Ο κύριος Καφ. Χθες άκουσα τον κύριο Μπαρνιέ να μιλάει για εύθραυστη ειρήνη. Αναφέρθηκε στο ότι συνάντησε οι γυναίκες που περνούν τα σύνορα στην Ιρλανδία για να πάνε στη δουλειά τους του είπαν ότι δεν θέλουν να, να υφίστανται ελέγχους. Εγώ ζητώ από τον κύριο Φαράζ και τους απέναντι να πάνε εκεί, να ακούσουν τις ιστορίες του κόσμου που ζει εκεί. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν πάντα εντάσεις. Η βία δεν είναι ποτέ μακριά. Οι Ιρλανδοί συνάδελφοι Μπέιλι και Μάρτιν έχουν άμεση πείρα από την κατάσταση των πραγμάτων προτείνουν μια ψηφοφορία για τους κατοίκους της Βόρειας Ιρλανδίας. Ας αποφασίσει η Βρετανική κυβέρνηση για τον backstop αφού ακούσει την άποψη των κατοίκων της περιοχής. Πιστεύουμε στα θαύματα, πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στην απέναντι πλευρά, πρέπει να πιστεύουμε στα θαύματα και δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας ότι θα υπάρξει μια λύση. Ευχαριστώ κύριε Κόφ και χαίρομαι για το ποίημα το οποίο επιλέξατε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγοντας τους συναδέλφους μέχρι τώρα στην Ολομέλεια κατάλαβα ότι η βασική ανησυχία είναι να ζητήσουμε την επανάληψη του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι ότου το αποτέλεσμα μας αρέσει, είναι αρεστώ σε μας. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία και θυμάμαι τι έγινε ε, όταν ε, εξελέγει η κυρία Φόντερ Λάιεν με εννέα ψήφους μόνο περιθώριο. Κανένας δεν ζήτησε να ξαναγίνει η ψηφοφορία. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να σεβαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί τότε αν ε, διαρρήξουμε τις σχέσεις μας σε ποιους θα πουλάμε τα γεωργικά μας προϊόντα, τα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προβλεπτικοί και όταν αποφασίσαμε να στηρίξουμε ε, το πιστοτικό σύστημα έγιναν ε, τεράστιες διάρκεια συνεδριάσεις, νυκτερινές ακόμα, για να στηρίξουμε τις τράπεζες γιατί δεν κάνουμε το ίδιο και για να στηρίξουμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Τσαμπάσκι, ένα λεπτό. Είναι προφανές όλο και περισσότερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός συμφωνίας και αυτό είναι εις βάρος όλων. Θα επηρεαστούν και οι εμπορικές συναλλαγές, θα τεθεί σε αμφισβήτηση η ειρήνη στην Ιρλανδία. Βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ και ένας από τους σημαντικούς εμπορικούς μας εταίρους. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για το προβλήματα στην Ιρλανδία και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κατανοήσουν ότι το backstop όπως το προτείνει ο κ. Μπαρνιέ δεν μπορεί να γίνει δεκτό ε, από τους Βρετανούς εταίρους μας. Εμείς μπορούμε να ελπίζουμε για μια σωστή συμφωνία όταν επιληθεί το θέμα του backstop. Αλλιώς θα θέσουμε σε κίνδυνο όχι μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την εμπιστοσύνη των βασικών μας εταίρων. Η κυρία Ροντρίγκε, ευχαριστώ πολύ. Για την Ισπανία είναι ένα μεταβατικό στάδιο το Brexit που δεν είναι καθόλου καλός ιονός. Μάλλον το Γιβραλτάρ θα ε, καταστραφεί και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ ε, και Ισπανίας. Μία ανοιχτή πληγή, 28.000 άνθρωποι περνάνε τα σύνορα κάθε μέρα, 13 από αυτούς δουλεύουν από την άλλη πλευρά. Δεν έχουμε καμία συμφωνία σχετική, ούτε οικονομική ούτε πολιτική. Τι θα γίνει με τις άδειες διαμονής, με τις άδειες εργασίας, τι θα γίνει με τις συντάξεις, με τις κοινωνικές εισφορές, με την οικονομική περίθαλψη που τους οφείλουν. Εάν φύγει χωρίς συμφωνία ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, τέσσερι ώρε ουρέ θα έχουμε στα σύνορα. Δεν θα έχουν τρόφιμα, δεν θα έχουν πρώτε ύλε. Τι θα γίνει με τι αγωγέ, εξαγωγέ και τον τουρισμό. Αυτό ο δρόμο στρωμένο ροδοπέταλα που φαντασιώνεται ο Τζόνσον θα είναι αδιαπέραστο με εκατομμύρια άτομα να κάνουν ουρά. Αν το κάνετε λοιπόν, αν θέλετε να φύγετε, αναλάβετε τις ευθύνες σας και μην παίζετε στα χαρτιά τις τύχες των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πώς σας πιέζω όλους με το χρόνο, αλλά σας παρακαλώ πολύ να μιλάτε πιο αργά, γιατί οι διερμηνείς ε, πρέπει να σας παρακολουθούν. Να λέτε λοιπόν λιγότερα στο χρόνο που σας δίνω. Επόμενος ο μιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Φόρμαν. Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη μου ομιλία στο Ευγενές αυτό κοινοβούλιο και ελπίζω και η τελευταία. Όταν μπήκα σε αυτό το κτίριο για πρώτη φορά είδα τεράστιε ταμπέλε. Μια τεράστια ταμπέλα που μιλούσε για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Αλλά γιατί να γίνονται δίκαιες εκλογές αν δεν τηρείται το αποτέλεσμα των εκλογών τι νόημα έχει να κάνουμε εκλογέ, αν αυτοί που έχουν χάσει δεν θέλουν να δεχθούν ότι έχασαν. Γιατί να έχουμε ελεύθερες και δίκαιε εκλογές αν θυσιάζεται η δικαιοσύνη των εκλογών γιατί η ελίτ πιστεύει ότι ξέρει ε, ε, ότι ε, καλύτερα από αυτού που ψήφισαν. Γιατί να μιλάμε για δημοκρατία στους καταπιεσμένους λαούς όταν δεν τηρούμε τα, αυτά τα οποία δημοκρατικά ε, ψήφισαν ε, οι λαοί των ίδιων των χωρών. αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει πραγματικά στη δημοκρατία, σε περίπτωση που ο Μπόρι Τζόνσον ζητήσει παράταση, θα πρέπει να απορρίψει το αίτημα. Αν πιστεύετε στη δημοκρατία, πρέπει ε, να υποστηρίξετε το λαό που ψήφισε στο δημοψήφισμα. Ζήτω συγγνώμη που διακόπτω την πρώτη ομιλία σας στο Κοινοβούλιο, λέει η Πρόεδρος, αλλά ξεπεράσατε το χρόνο σας. Κύριος Μπέλαμι, μισή λεπτό. Derrière les éclats. Πίσω από τις φωνές που ακούμε σήμερα το πρωί υπάρχουν σαφείς κινδυνοί για τις χώρες μας. Ο λαός της Βρετανίας επέλεξε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γίνει σεβαστή επιλογή του. Αλλά ο σημερινός διάλογος είναι χρήσιμος όχι μόνο για να κρίνουμε την πολιτική ζωή της Βρετανίας αλλά και για μας, όπως υπενθυμίσατε κύριοι διαπραγματευτές, πρέπει και για μας να είναι σημαντική η προστασία όλων των πολιτών θα είμαστε όλοι περισσότερο ευάλωτοι εάν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερο ευάλωτοι έναντι ε, των απειλών ε, και είναι σημαντικό στοιχείο για τις ε, δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα είμαστε περισσότερο αδύναμοι έναντι της τρομοκρατικής απειλής ή όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα. Είναι γενικά δύσκολο το γενικό πλαίσιο και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο σημαντικό πλήγμα μιας αποχώρησης χωρίς συμφωνία για τις γειτονικές χώρες μεταξύ των οποίων τη Γαλλία που σε περίπτωση αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να διαχειριστεί το βάρος ε, ε, ε, των συνόρων με την Μεγάλη Βρετανία. Ιδιαίτερα στον τομέα της αλίας, διότι το κλείσιμο της Βρετανίας θα είναι τεράστιο πλήγμα και για τους δύο. Περιμένουν από εμά χιλιάδες πολιτών, εκατομμύρια πολιτών να είμαστε υπεύθυνοι δεν είμαστε εδώ για να ξαναρχίσουμε ένα δημοψήφισμα στο οποίο ήδη έχουν ψηφίσει οι πολίτες, αλλά για να βρούμε μια συμφωνία. Και ελπίζουμε, αγαπητέ Μισελ, ότι θα φροντίσετε να έχουμε μια σωστή συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκυγιόμ, ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Και επίσης υπάρχουν ανησυχίε για τη συμπεριφορά του Βρετανικού Πρωθυπουργού. Μέσω του ψηφίσματος εμείς εδώ προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους Βρετανούς. Θέλουμε μια συντεταγμένη αποχώρηση με εξασφάλιση της ειρήνης στο, ε, στο, ε, στην Ιρλανδία και με μια ε, τακτική ρύθμιση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στη Βρετανία και αντιστρόφως. Εκεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και τις διατάξεις για τα διαζύγια. Τώρα λοιπόν περιμένουμε με ανησυχία τι θα πει ο Βρετανός Πρωθυπουργό. Περιμένουμε τις ε, προτάσεις που θα καταθέσει, που θα είναι ε, εύκολο να τις κατανοήσουμε και όπου θα αναλαμβάνει τις υποχρεώτες τους. Γιατί εδώ και τρία χρόνια μας είπανε ε, ε, πως ο Ντέιβιτ Κάμερον το είπε στον τύπο πως εδώ και τρία χρόνια ε, σιωπηλά ε, βασανίζεται γιατί δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα του μετά από την απόφαση που πήρε να κάνει δημοψήφισμα. Ανησυχούμε κι εμείς. Ο κύριος Καρικάνο πάνω από 50.000 Ισπανοί ζουν στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από 300.000 Βρετανίζουν στην Ισπανία. Αυτό το καθαρό Brexit που αναφέρει ο κ. Φάραντζ για μας είναι πολύ βρώμικο. Και η κατάσταση είναι δραματική. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στο Ηνωμένο Βασίλειο και συζητούσα εκεί με Ισπανούς πολίτες. Ανησυχούν γιατί ε, έχουν αυτό το καθεστώς του ε, μακροπρόθεσμα διαμένοντα ε, και είναι τελείως ασταθές ε, και δεν ξέρουν τι θα συμβεί αν ο κύριος Φάρατ και ο κύριος Τζόνσον συνεχίσουν με την τακτική της μιλήσης. Φανταστείτε τι ζουν αυτοί οι πολίτες μας, οι οποίοι μετά από δεκαετίες ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν τη βεβαιότητα αν οι ζωές τους μπορεί να συνεχίσουν εκεί ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσει τους πολίτες της το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κάνει το αντίστοιχο. Θα πρέπει εμείς λοιπόν να τους στηρίξουμε και θα πρέπει να αποφύγουμε την άτακτη αποχώρηση το Brexit χωρίς συμφωνία που θα ήταν καταστροφικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό η κυρία Ρέντκε. Ας είμαστε ειλικρινοί συνάδελφοι πολύ κουράστηκαν, πολύ εξαντλήθηκαν, πολλοί θέλουν να προχωρήσουν. Πιστεύουν πως αν δεν δώσουμε την επέκταση προθεσμίας θα συνεχίσουμε κάνοντας τα υπόλοιπα που χρειάζεται να κάνουμε και όλα αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν τους τελευταίους μήνες και χρόνια θα τα αφήσουμε πίσω μας. Συνάδελφοι, μην κάνετε το λάθος αυτό. Εάν δεν δοθεί αυτή η παράταση, εάν δεν αποφύγουμε το Brexit χωρίς συμφωνία, ο εφιάλτης δεν θα τελειώσει. Τα σύνορα μεταξύ ΙΡΕ και Βορείου Ολλανδία δεν θα λυθούν. Τα δημοσιονομικά δεν θα λυθούν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, το μέλλον αυτών, δεν θα λυθούν. Συνάδελφοι, δεν είναι η στιγμή τώρα για να φωνούμε κοντόφθαλμοι. Αντίθετα, για να προσφέρουμε αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη με τις εκατοντάδες χιλιάδες ε, πολιτών των Ηνωμένων Βασιλείων που κάνουν πορείες, διαμαρτυρίες και καλούν εμάς να τους χορηγήσουμε αυτή την παράταση για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο, να βρεθούμε μια λύση ε, για αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι σε εσά θα δώσω το βραβείο για το σεβασμό του χρόνου που σας είχε δοθεί ο μιλητής και δεν θέλω να σας πιέσω, κύριε Κρασναντέψη, αλλά έχετε ένα λεπτό στη διαθέσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω τη συζήτηση αυτή και θέτω το ερώτημα ποιο είναι το συμπέρασμα από μια τέτοια συνάντηση, τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι το συμπέρασμα είναι το εξής θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα, για το χειρότερο σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται κανείς δεν το θέλει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτό το σενάριο φαίνεται να προχωρεί προς υλοποίηση. Και θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα για το μέλλον, υπευθυνότητα για τις καταστροφές που θα επέλθουν. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύτέ μας και ο κύριος Μπαχνιέ και ο κύριος Γιούνκερ το καταλαβαίνει αυτό, καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την καταστροφή όσο είναι δυνατόν. Αναβάλλοντας το Brexit επάπειρον δεν θα οδηγήσει πουθενά, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο χάος και αβεβαιότητα. Παρακαλώ λοιπόν να αναλάβετε δράση. Ευχαριστούμε. μισή λεπτό, κύριος Άγγελ. Είναι προφανές ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Λυπούμεθα γι' αυτό, αλλά σεβόμαστε την επιλογή του Βρετανικού λαού. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν με ένα πραγματικό πνεύμα καλής πίστης και συνεργασίας για να βρεθεί καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές. όλα αυτά οφείλονται στην ε, σταθερότητα και στην ε, γαλήνη που έχει επιδείξει ο Μισελ Μπαρνιέ ε, και στην καλή πίστη που έχει επιδείξει. Και γι' αυτό αν ε, κανένας πολιτικός ηγέτης δεν σέβεται την Βρετανική θέση, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα λύπηρο. Είμαστε δυνατοί λοιπόν, συνεχίζουμε Είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε το αίτημά σας για παράταση αν είναι τεκμηριωμένοι. Ε, μπορείτε να υπολογίζετε σε μας αλλά αναμένουμε και αμοιβαιότητα. Είναι καιρός να πιεστεί ο κύριο Τζόνσον. Είναι λυπηρό που εσείς χρησιμοποιείτε Αμερικανούς υπερίοες ε, των κινούμενων σκίτσων. Έχετε καλύτερες πηγές έμπνευσης στην λαϊκή σας παράδοση. Κύριε Τζόνσον, πιστεύετε ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ο Incredible Hulk ή μήπως οι δυνατότητες του Χάρι Πότερ και οι μαγικές του ιδιότητες. Ξεχάστε τον Αμερικανό Χάλτ. Λοιπόν, πρέπει να, είμαι, να αντιμετωπίζω όλο τον κόσμο ισότιμα, δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Ράντσελ, ε, θα έχετε το λόγο αν δέχεστε την ερώτηση από τον κύριο Χάπεμπ. 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση και 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Χάμπιμπ. Για τρία χρόνια ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κανόνες. Ο κύριος Ράγκελ αναφέρθηκε στην διάθεση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσει μαζί μας και τα θέματα του backstop. Να θυμίσω όμως ότι ε, στη συμφωνία ε, για την παράταση μετά τις 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης. Δεν θα σας ζητήσω ε, να απαντήσετε στην ερώτηση διότι ε, ακολούθησε τα 30 δευτερόλεπτα. Μορένο Σάντσες. το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει, φαίνεται, θα οδηγηθεί φαίνεται σε ένα σκληρό Brexit σαν αποτέλεσμα ε, των ανεύθυνων πολιτικών, των πολιτικών ηγετών που θα οδηγήσει σε προβλήματα και τον λαό της χώρας και που έκλεισε και το ε, Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια ιστορική ε, στιγμή και η στάση των Ισπανών Σοσιαλιστών είναι σαφής και συμβατή με το ψήφισμα που έχουμε ε, σήμερα να ψηφίσουμε. Όχι στο σκληρό ε, Brexit, ναι σε μια συντεταγμένη αποχώρηση. Μια μη συντεταγμένη αποχώρηση δεν θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών μας. Μια συμφωνία όμως που θα προστατεύσει μέσω του backstop την ειρήνη ε, στην ε, Ιρλανδία και θα διατηρήσει και την ακαιρεότητα της εσωτερικής ε, αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καθυστερήσει. Θα πρέπει να προχωρήσει και η Βρετανική κυβέρνηση. Για ένα λεπτό, κυρία Μπέα πρόεδρε, συνάδελφοι, το σενάριο της αποχώρησης χωρίς ε, συμφωνία είναι σαφές. Όλοι γνωρίζουμε τις καταστροφικές συνέπειες, ιδιαίτερα για τους πολίτες ε, της Ιρλανδίας και των υπεράκτιων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προσπάθεια για τα μέτρα, ε, αν θέλετε, τα διορθωτικά προχωράει γρήγορα ιδιαίτερα να δούμε τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης να συγχαρώ και τους συναδέλφους ε, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που θέλουν να βάλουν στη θέση του τον ε, Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτό θα οδηγήσει σε μια παράταση έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία ή και σε μια δεύτερη ευκαιρία εν πάση περιπτώσει ελπίζω ο Θεός να προστατεύσει την τύχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κύριος Μπιτό ένα λεπτό. Πρόεδρε, η υπόθεση μιας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία ε, είναι κάτι το πολύ πιθανό πια. Και γι' αυτό οι συνέπειες στη Γεωργία και την Αλληλεία θα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές. Ε, στο βόιο κρέας, ε, στην τυροκομεία, ε, επίσης στα ποτά. Η κρίση θα είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς προχωράμε χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί. Οι Ιρλανδοί παραγωγή βοήου κρέατος, όπως είπε ο Φλάναγκαν, αντιμετωπίζουν τραυματικά προβλήματα. Προσπαθούν να βοηθηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι ανησυχίες τις οποίες έχει εκφράσει ο Φιλ Χόγκαν είναι βάσιμες. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε όλους τους Ευρωπαίους αγρότες που θα επηρεαστούν αρνητικά από το άτακτο Brexit. Η κυρία Βετσόνοβα. Το Brexit έρχεται σε λιγότερο από 1,5 μήνα έρχεται το Brexit ε, και θα πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ακόμη και αν δεν το επιθυμούμε. Πολλοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της άμεσης δημοκρατίας το δημοψήφισμα είναι η πιο καθαρή μορφή δημοκρατίας και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πρέπει να γίνει σεβαστό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον εναπομένοντα χρόνο για να εμποδίσουν ένα σκληρό Brexit, το οποίο θα είναι επιζήμιο όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Για να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία χρειάζεται έγκριση και από τους δύο συμβαλωμένους. Είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμφωνεί με την τρέχουσα μορφή της συμφωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η συμφωνία. Ευχαριστώ η κυρία Ντελάνγκε. μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, ο λόγος για τον οποίο μπήκα στην πολιτική κάποτε ήταν η οθόδης πυρετός και ήταν μια ασθένεια των ζώων που δεν σταματάει στα σύνορα, δεν ξέρει σύνορα, δεν θα σταματήσει ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Θανατώθηκαν εκατομμύρια ζώα για μια ασθένεια που θα μπορούσε να είχε αποφευθεί με κατάλληλο εμβολιασμό. Και σε αγροτικές περιοχές η απογοήτευση που δημιουργήθηκε δεν έγινε είναι ακουστή στο Λονδίνο, γιατί δεν ήθελαν οι πολιτικοί εκείνη την εποχή να αλλάξουν την πολιτική του μη εμβολιασμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα και των Βρετανών πολιτών και των υπολείπων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυτό το οποίο ακολούθησε τη σωστή πολιτική. Είχα συνεργαστεί τότε ε, με όλους για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τις καταστροφικές συνέπειες ε, με εκπροσώπους ε, και των συντηρητικών και άλλων. Σήμερα το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει κλείσει, δεν λειτουργεί και μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε λειτουργία για να υπερασπίσει τα συμφέροντα και των Βρετανών και των υπολείπων Ευρωπαίων πολιτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει ε, μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία, αλλά δεν ε, ε, θα δεχθούμε να μην έχουμε εποπτεία των χρηματοοικονομικών προϊόντων, ούτε χαμηλά πρότυπα για το περιβάλλον. Και αν θέλετε το λόγο, ρωτήστε τους πολίτες και στο Northumberland, αλλά και στην, στο Friesland, στην Ολλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καμπούλενάτη. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, εκπροσωπούμε τους πολίτες από διάφορα κράτη-μέλη και θεωρούμε πολύ σοβαρό το θέμα του Brexit και γι' αυτό συμμετέχουμε θερμά σε αυτή την προσπάθεια με τους Βρετανούς συναδέλφους. Το Κοινοβούλιο είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. στο δυτικό πολιτισμό ε, το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε γιατί η συμφωνία έχει περάσει και από τις δύο βουλές του Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, τώρα φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ε, προσπαθεί να αφαιρέσει τον έλεγχο από το Κοινοβούλιο και από τους πολίτες η ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει να επιθυμεί το Brexit χωρίς συμφωνία και φαίνεται να ακολουθεί μια πιο σκληρή γραμμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρεμείνει λογική και ήρεμη. Να δώσουμε χρόνο στους Βρετανούς αν θέλουν να ξεκαθαρίσουν το χάος που έχουν δημιουργήσει. Η κυρία Χαραντζόβα, ένα λεπτό. paní Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμά δεν επιθυμούμε το Brexit. Πολλοί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να συμβεί το Brexit. Αλλά ο Βρετανός Πρωθυπουργό ε, είναι έτοιμος να τα καταστρέψει όλα, να φύγει χωρίς συμφωνία. Το, τη χειρότερη επιλογή. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να προετοιμάζεται ακόμη και για αυτό το χειρότερο σενάριο. Και επιπλέον η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Δεν θα πρέπει να τι αφήσουμε να καταρρεύσουν μαζί με το Brexit. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τους ε, πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν ε, στα νησιά του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς να ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν φαίνεται να ισχύει πια τίποτα. Ανατρέπονται οι συμφωνίες, αυτά τα οποία αναμένονταν δεν υλοποιούνται και χάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση την υπομονή της. Ευχαριστώ. κύριο Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να στραφώ προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας πω πως από τη συζήτηση προκύπτουν ε, τρία προβλήματα αν έχουμε άτακτη υποχώρηση. Πρώτα απ' όλα βεβαιότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί αν υπάρξει συμφωνία τα δικαιώματά τους εξασφαλίζονται. Δεύτερον, ένα έλλειμμα 50 περίπου δις ευρώ που είναι το ποσό το οποίο έχει αναλάβει ως ε, υποχρέωση ως δέσμευση πληρωμής στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο μέχρι το 2020. Και τρίτον, τα προβλήματα στο αμοιβαίο εμπόριο. Έχουμε μεγάλο πλεόνασμα ε, γύρω στα 100 δις ε, λίρες για το 2017 ε, με το εμπόριό μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και καταλαβαίνετε πως εάν δεν έχουμε συμφωνία οι εμπορικές συναλλαγές θα γίνονται σε καθεστώς ΠΟΕ με δασμούς και ποσοστώσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει πως θα βρούμε συμφωνία με μια τροποποιημένη πολιτική δήλωση και με κάποιες ε, χειρονομίες καλής βούλησης προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νίντε Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως τα πιο σημαντικά κομμάτια και σχόλια για το Brexit τα έχουν πει όλοι ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 27, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, ας μην χάσουμε την ευκαιρία να φτάσουμε σε συμφωνία. Μια συμφωνία που θα μειώσει το κόστος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για όλους τους Ευρωπαίους και για τους Βρετανούς και για ε, τους Βρετανούς που ζουν στην υπηρετική Ευρώπη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως η παράταση αυτή ε, να λύσει κάπως το πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να διδαχτούμε από τους φίλους στο Λονδίνο τι μπορεί να κάνουμε για να είναι η κοινωνία μας πιο δίκαιη και να αποφεύγουμε κρίσεις σαν αυτές που ζουν στο Λονδίνο. Καταρχήν, οι πολιτικοί θα έπρεπε καμιά φορά να παραδέχονται πως τα προσωπικά τους συμφέροντα, εξουσίες ή ε, νίκες, εκλογές για αυτούς έχω μεγαλύτερη σημασία από το τι θα συμβεί στη χώρα και στην κοινωνία. Και δεύτερον, και όχι μόνο για τους πολιτικούς, θα πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας όταν οι απόψεις μας αποκλίνουν. Καλύτερα να οικοδομούμε γέφυρες και όχι τείχη. Και τέλος, θα πρέπει να προωθήσουμε την εξής νοοτροπία. Πως η αλήθεια θα πρέπει να πριτανεύει και να μην προωθούμε το ψέμα. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως αυτές οι ανησυχητικές τάσεις που έχουμε στις κοινωνίες μας, όπου επιβραβεύεται το ψέμα και όχι η αλήθεια, θα ανατραπούν και θα αντιστραφούν και πως οι μεγαλύτεροι ψεύτες δεν θα γίνονται ούτε πρωθυπουργοί ούτε πρόεδροι. Για ένα λεπτό ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, θα ήθελα να συμπισήσω την προσοχή στο εξή. Πολιτική υπευθυνότητα για την τύχη της Ευρώπης. Και αυτή η πολιτική υπευθυνότητα είναι μια αρχή η οποία θα πρέπει να διέπει τις σκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάνω από ένα εκατομμύριο Πολωνοί ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσπαθούμε το εμπόριο, το βιομηχανία μας, τις μεταφορές, τα οικονομικά μας σημεία να τα προστατεύσουμε. Όμως η έλλειψη υπευθυνότητα χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχω την εντύπωση πως ε, θεωρεί πως όλα είναι ευθύνη δική μας η, του Ηνωμένου Θέλουν μόνο τα πλεονεκτήματα και δεν θέλουν καθόλου να μοιραστούν την ευθύνη για τα μειονεκτήματα της απόφασής τους. Και δεν βλέπω καμία επικοδομητική πρόταση ως προς ενδεχόμενες λύσεις. Ή θα γίνει, θα συνεχίσει η ζωή και μετά τον Brexit, οπότε χρειαζόμαστε αμοιβαία εμπιστοσύνη και ζητώ από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να οικοδομήσει αυτή την εμπιστοσύνη, γιατί διαφορετικά καλή λύση δεν θα βρούμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κιουτσούκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Τρία χρόνια μετά την απόφαση ε, του Βρετανικού λαού ε, λαμβάνουμε ένα μήνυμα ισχυρό. Ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν είναι ο εκφραστής του Βρετανικού λαού, δεν είναι η φωνή του. Κάθε μέρα μας στέλνουν μηνύματα κατά το Brexit. Και έχουμε τόσους πολλούς ε, Βρετανούς ε, ευρωβουλευτές που είναι υπέρ της παραμονής. Τώρα χρειάζεται μια αλλαγή, γιατί το Brexit το επιδιώκουν για τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στο κόμμα των συντηρητικών. Αλλά δεν ξέρουν πώς θα το εφαρμόσουν. Επιμένουν να αφαιρέσουμε το backstop. Αλλά δεν προτείνουν κάποια λύση που να λειτουργεί. Η Βρετανική κυβέρνηση λοιπόν δεν προσπαθεί να πετύχει μια συντεταγμένη αποχώρηση. Τα παιδιά σας, οι φοιτητέ σας, οι δικοί μας πολίτες χρειάζονται βεβαιότητα. Πάνω από 3 εκατομμύρια ε, Βρετανοί ε, δεν είναι Βρετανοί πολίτε, αλλά είναι, για παράδειγμα, πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλοί από τη δική μου χώρα, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή του και την ανησυχία του μετά το δημοψήφισμα. Είναι κακή ιδέα το Brexit και θα πρέπει να σταματήσει πια. Uh, λεπτό, eh, er Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά ακούστηκαν. Αυτό το οποίο είναι όμως σαφές είναι ότι το Brexit αντιπροσωπεύει μια τεράστια πρόκληση και η έλλειψη συμφωνίας θα θέσει σε κίνδυνο 1.250.000 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στο Βέλγιο θα απολεσθούν τουλάχιστον 30.000 ε, θέσεις. Η επιλογή της Βρετανικής κυβέρνησης δεν είναι σαφής, η αβεβαιότητα αυξάνεται και κανονικά θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια συμφωνία προς το συμφέρον του λαού της Ευρώπης και των επιχειρησιών της. Είναι σαφές ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να προστατευτούν επαρκώς κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Πρέπει και το Βρετανικό Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθεί τάχιστα έτσι ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας. Το Brexit ε, έχει συζητηθεί πάρα πολύ μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων δυστυχώς δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Και έχουμε μια εθνική διαφορά, εσωτερική διαφορά σε μια χώρα που επηρεάζει όλη την Ευρώπη. ο κύριος Μπαρνιέ και η ομάδα του κατάφερε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις αλλά δυστυχώς η κατάσταση στην άλλη πλευρά της μάχης είναι χαοτική και έχουμε και ένα κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ ε, ε, μεγάλες πιέσεις και είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς σήμερα τι ανήκει σε στρατηγική επιλογή, τι είναι μπλόφα και θα πρέπει σε καμία περίπτωση η ενότητα της Ένωσης να αμφισβητηθεί μέσω του Brexit. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπίλτσικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πολίτες είναι, αν θέλετε, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής μας λειτουργίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υποστήριξε τους διαπραγματευτές για τον Brexit γιατί είναι σημαντικό για τις ζωές των πολιτών. Το ψήφισμα εμένει στην ενότητα των 27. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα είναι να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση για να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από μικρές και μεγάλες χώρες. Πρέπει ε, σε, ε, σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς καθυστερήσεις και παλινοδίες, να προσφέρει η Βρετανική κυβέρνηση την μόνιμη δυνατότητα παραμονής ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του Brexit με ενότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ενοποιημένα το χειρότερο σενάριο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ενότητα των 27 ήταν, ε, θα έλεγα, ο πυρήνας της διαπραγματευτικής ικανότητάς μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί. Ρέγνα. Ευχαριστώ. Εδώ και τρία χρόνια οι σκληροπυρηνικοί του Brexit δεν έχουν κανένα σχέδιο για το πώς θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουν ε, ε, ότι μπορεί να σωθούν και με μία έξοδο χωρίς συμφωνία, κάτι εναντίον του οποίου έχουμε προειδοποιήσει πολλές φορές ότι δεν πρέπει να συμβεί. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, τα δικαιώματα των γυναικών εργαζομένων, των παιδιών, της μητρότητας. Όλα αυτά μπορεί να χαθούν με ένα σκληρό Brexit κυρίως ε, οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προστατευθούν γιατί πολύ συχνά ε, απασχολούνται σε τομείς όπως το εμπόριο ε, ή στον τομέα της υγείας και πρέπει να ενισχυθούν οι κοινωνικές τους παροχές. Όσο μπορούμε να τίνουμε χείρα βοηθείας προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε πάντοτε είναι προτιμότερη στάση έναντι του να πούμε ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ο κύριος Κίρτσος, ένα λεπτό. Νομίζω ότι το θρίλερ του Brexit έχει κοινά σημεία με το θρίλερ του Grexit το 2015. Και ο Μπόρις Τζόνσον, αν και είναι τελείως διαφορετικός από πολιτική άποψη, έχει κοινά σημεία στην τακτική του με τον Αλέξη Τσίπρα. Και οι δύο έβαλαν το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό συμφέρον και οι δύο για ένα διάστημα υποκρίθηκαν ότι διαπραγματεύονταν ενώ ουσιαστικά πηγαινοέρχονταν στις πρωτεύουσες. και οι δύο υποκρίθηκαν ότι δεν τους ενδιέφεραν οι συνέπειες των πράξεών τους και ότι δεν είχαν έτσι αίσθηση του ρίσκου. Ο Τσίπρας όμως προς τιμήν του έκανε την τελευταία έστω στιγμή μια στροφή 180 μοιρών πιεζόμενος από εμάς, πιεζόμενος από τη σκληρή πραγματικότητα και βοηθούμενος από τον πρόεδρο Γιούνκερ δυστυχώς δεν νομίζω ότι ο κύριος τζόνσον θα ακολουθήσει το καλό παράδειγμα του τσίπρα και, δεν θα, πιστεύω δεν θα βελτιώσει την πολιτική του. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να παρακολουθούμε το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το Βρετανικό λαό, τη Βρετανική νεολαία και να του στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε μαζί τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαλντεμόζε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θεωρώ λυπηρό. Αυτή όμως αποτελεί και την επιλογή των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να το σεβαστούμε. Όμως, είναι σχεδόν αδύνατο να συγχωρήσουμε την επιλογή η αποχώρηση να γίνει μέσω σκληρού Brexit. Θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για τεράστιο αριθμό ανθρώπων από την άλλη πλευρά της μάχης. Ε, το κόστος θα είναι θέση εργασίας, θα επηρεάσει τους φοιτητές, τους ερευνητές. Νομίζω πως είναι απαραίτητο να δώσουμε λίγο χρόνο έτσι ώστε να αποφύγουμε το σκληρό Brexit και να μην επηρεαστούμε τον τρόπο αυτό οι οικονομίε μα και οι πολίτε μα. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζω και εγώ στο να παρατείνουμε λίγο το χρόνο για να βρούμε μια συμφωνία. Α αποφύγουμε το σκληρό Brexit. Δεν ε, συμφέρει κανέναν. Ο κύριο Warborn, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να πω δύο λόγια για το Brexit. Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις εμπορικές σχέσεις. Ε, για ε, τη Σουηδία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος, αλλά βέβαια το εμπόριο δημιουργεί θέσεις εργασίας και φροντίζει για την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit είναι κίνδυνος και για τις θέσεις απασχόλησης. Χαίρομαι γιατί στο ψήφισμα υπάρχει δυνατότητα για παράταση της προθεσμίας. Παράταση μέχρι ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να δώσουμε ε, γενναιόδορες ε, δυνατότητες για τον Brexit σε περίπτωση που ζητηθεί από τους Βρετανούς ε, μια παράταση και να μην ε, αγνοήσουμε τη σημασία που έχουν οι εμπορικές συνθήκες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φχίτζον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σε λίγες εβδομάδες ε, μπορεί, λόγω του Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το συμφέρον όλων των πολιτών και για τους πολίτες βέβαια και για τις επιχειρήσεις θα είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες. Στη Σουηδία είναι πολλοί οι πολίτες που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σκέφτονται να αποχωρήσουν ή έχουν ήδη αποχωρήσει. Αβεβαιότητα για το μέλλον υπάρχει και για τους Βρετανούς. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ισορροπημένο και προτείνει αυτά τα οποία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές για μια πιθανή αποχώρηση. Θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία με διαφάνεια για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. και από τον κύριο Τζόνσον ζητώ να φροντίσει το μέλλον της χώρας του. Ευχαριστώ. Κύριος Μακάλιστερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να τονίσω πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν και από τους συναδέλφους σήμερα το πρωί, αλλά να προσθέσω και μία διάσταση στο Brexit χωρίς συμφωνία σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Ο Μισελ Μπαγνιά αναφέρθηκε στην πολιτική διακήρυξη. Ναι, η πολιτική διακήρυξη, στην οποία συμφώνησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβάνει δικαστική αστυνομική συνεργασία, νευρή χώρο δικαιοσύνη. Ε, εξωτερική ασφάλεια και άμυνα. Με ένα Brexit χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορεί πλέον να συνεργάζεται σε υφιστάμενα και μελλοντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και στην ΚΕΠΑ. Και δεν θα μπορούν ε, και, ευρωπαϊκές, και βρετανικές εταιρείες να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά έργα. Αυτά είναι επιχειρήματα προς τους συναδέλφους της ακροδεξιάς ε, που δείχνουν πόσο είναι σημαντικό να αποφύγουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία ε, με κάθε δυνατότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους ε, που προετοίμασαν ε, το ψήφισμα το οποίο θα υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Α είμαστε ξεκάθαροι ποιο φταίει για αυτό το χάο. Ξεκινά κανεί με υποσχέσει που δεν μπορεί να υλοποιήσει, λέγοντα ότι θα κρατήσει ε, ε, τι υφιστάμενε σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιο θετικά. Μετά ε, λένε ότι είναι σε θέση ισχύω φεύγοντα από ένα τόσο ισχυρό όμιλο κρατών και στη συνέχεια καταλήγουμε να βλέπουμε ότι ακόμη και στα έγγραφα της χώρας ε, υπάρχουν προβλέψεις ε, για ελλείμματα φαρμάκων που θα απειλήσουν τους πολίτες της χώρας σε περίπτωση του Brexit. Ε, κύριε Μπαχνιέ, θέλετε να προχωρήσετε. Όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε και ξέρω ότι πολλοί από τους συναδέλφους μου έχουν βαρεθεί αυτό, αυτή την κατάσταση. Το καταλαβαίνω. Αλλά ας μην προσποιούμεθα ότι χωρίς να το εγκρίνει ο λαός θα είναι επιτυχημένο το Brexit. Θα πρέπει ε, ο λαός της Βρετανίας να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το κατά πόσο θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Δώστε μας τη δυνατότητα να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε ένα Να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κύριο Μπαρνιέ για την επαγγελματικότητα που επέδειξε. Στην ουσία είχαν πει οι οπαδοί του Brexit ότι θα απαλλαγούν από ένα πτώμα, θα ξεφύγουν από το πτώμα στο οποίο ήταν προσδεδεμένοι. Εμείς φαίνεται ότι σαν πτώμα είμαστε πολύ ζωηροί και εξακολουθούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας όπως για την μη ύπαρξη σκληρών συνόρων στην Ιρλανδία όπως και για το backstop ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ανεξαρτήτως αυτών που γίνονται ή δεν γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Άγγλοι υπερεθνικιστές είναι οι υπέρ της έλλειψης συμφωνίας. Η κυβέρνησή σας λέει ότι θα ήταν καταστροφή. Να ρωτήσω από τον κύριο Φαράζ και τους συνενόχους του το εξής. Αν τα καταφέρετε και αν πράγματι η Βρετανική κυβέρνηση είναι σωστή για τις συνέπειες της μη συμφωνίας, μη μας κατηγορήσετε για τις συνέπειες. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την βοήθειά σας στο σεβασμό του χρόνου. ένα λεπτό. ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και 70 χρόνια εμείς αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την πολιτική μας ένωση. Το κάναμε αυτό γιατί γνωρίζαμε ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε κάθε χώρα. Δυστυχώς το 2016 με το δημοψήφισμα του Brexit μια μικρή πλειοψηφία αποφάσισε την αποχώρηση. Τότε είχαμε πει ότι ήταν η υπαρξιακή κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η υπαρξιακή κρίση δεν είναι στην Ένωση, είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Ο κύριος Τζόνσον είναι σε θέση να σεβαστεί ε, τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει μετά από την ψηφοφορία της κάτω βουλής. Αν δεν το κάνει οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Φιτζέραλτ. Πολύ ξεχνάτε και κάποιοι αγνοείτε το γεγονός που πίσω από τα πολιτικά σλόγγαν και τις δηλώσεις κρύβονται πραγματικοί άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, των οποίων οι επιχειρήσεων και η ασφάλεια κινδυνεύουν. Η ειρήνη επίση πάνω στις οποίε αυτές οι ζωές έχουν οικοδομηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η δημοκρατία από την πρώτη μέρα απερίφραστα είπε πως θα κάνει αποφασιστικά ό,τι χρειάζεται με ή χωρίς συμφωνία για να αποφύγει την ανάγκη συνόρων και να εξασφαλίσει την ειρηνευτική διαδικασία. Είναι μια διεθνή συμφωνία με εγγυήτριες δυνάμεις. Μην το ξεχνάτε. Οποιοδήποτε επιπρόσθετες ιδέες κατατεθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο θα, θα ε, τύχουν πολύ θετική υποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ε, εξεταστούν. Αλλά εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτούμε οποιαδήποτε συμφωνία που να μην εξασφαλίζει ε, αυτά τα οποία έχουμε μέσα στο backstop, που είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή στο τραπέζι που αποφεύγει ο, οποιαδήποτε φυσική υποδομή μεταξύ των συνόρων. Όπως είχε πει και ο Τζον Χιούμ, όταν ο κόσμος ε, είναι διαιρεμένος, η μόνη λύση είναι να τον κάνει να συμφωνήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω 19 αιτήματα, θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τους ε, πέντε, αλλά νομίζω ότι θα απογοητεύσετε κάπως, γιατί κάποιοι δεν θα προλάβουν. Η κυρία Σόιτροβα να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι γνωρίζουμε πως το Brexit θα αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο θα αποδυναμώσει και το Ενωμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον κύριο Φάραντζ. Πώς μπορείτε να λέτε πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι δυνατότερο ίσως πιο δυνατό από τις μικρές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν έρθετε να αντιμετωπίσετε τη ΣΥΠΑ, την Ρωσία, την Κίνα, δεν θα είστε σε καλύτερη, θα είστε ο πιο αδύναμος. Και γι' αυτό λυπάμαι για τη θέση σας και για την πολιτική επιλογή που κάνατε. Όταν οι ψηφοφόροι σας επέλεξαν, δεν επέλεξαν ψηφίζοντας το χάος αυτή την ε, αποχώρηση χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η θέση τους πια θα είναι ασταθής. Βέβαια, αν φύγετε χωρίς συμφωνία και πάλι θα πρέπει να διαπραγματευτείτε μια νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για να συμβεί αυτό Λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις προϋποθέσεις που θα σας θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας παρακαλώ πολύ. Η κυρία Ward για ένα λεπτό. Με την Πρωθυπουργία Τζόνσον εμείς είμαστε μάρτυρες στο ότι η αξιοπρέπεια υποχωρεί την εποχή του λαϊκισμού. Ο Τζόνσον είναι ο πιο κακόφημος Πρωθυπουργό, είναι ντροπή για το κόμμα του και για τη χώρα του. Ε, μισογίνης, Ισλαμόφοβος, ε, ομόφοβος, επικίνδυνος κλόουν, τον οποίο επέλεξε κάτω από 2% του πληθυσμού μας έχει κάνει ό,τι να είναι με τις ζωές των ανθρώπων και το Brexit χωρίς συμφωνία ε, έχει τον κίνδυνο του να λείψουν τα απαραίτητα φάρμακα και τρόφιμα. Απειλεί την συμβίωση σε ειρήνη. Ναι, όχι μόνο λοιπόν δουλειές αλλά και ζωές θα χαθούν από τον Brexit αυτού του είδους και η κυβερνητική πολιτική αποφασίζεται από έναν μη ε, ερετό ε, σύμβουλο, τον ε, Dominic Cumming, ο οποίος αυτή τη στιγμή περιφρονεί το κοινοβουλίο του. Έτσι έχουμε ξαναναλάβει τον έλεγχο. Έχω μια κυβέρνηση που καταστρέφει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς του. Σας ευχαριστώ πολύ, Τζούλια. Έληξε ο χρόνος σου. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρο, αλλά αν όλοι ξεπερνάνε το χρόνο, λιγότεροι ομιλητέ θα μπορέσουν να μιλήσουν. Ο κύριο Νιούτον Ντάν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προ τον Επίτροπο Μπαχνιέ. Δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει μετά από τη συζήτηση αυτή. Πολύ απλά. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, ισχύει ότι οι ανταλλαγέ πληροφοριών μεταξύ Europol και αστυνομικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα διακοπούν. Επομένω, η δυνατότητα αντιμετώπιση ε, της εγκληματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα είναι πολύ χαμηλότερε. Thank you. Colleagues, I want to start by apologizing for the behavior of a small minority of my compatriots. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για τη μειονότητα των συμπολιτών μου και στο Κοινοβούλιο και στη χώρα μου που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς να αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία στη χώρα μου, λέει η κυρία Τσόνς. Ε, το Brexit δημιουργήθηκε από αυτού οι οποίοι θέλουν την αποχώρηση, γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για το τι είδο Brexit θα ήθελαν. Λόγω Τη εσωτερική κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε ψήφο για το λαό για να μπορέσουν να επιλέξουν οι πολίτε ανάμεσα σε μια σαφή επιλογή για την αποχώρηση και ε, την παραμονή από την άλλη πλευρά που είναι για μας η καλύτερη λύση. Η αποχώρηση χωρίς συμφωνία δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Είναι αυτοκαταστροφική και επιζήμια. Σας παρακαλώ συνάδελφοι, κάνετε ό,τι μπορείτε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε μέρα στους δρόμους και στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζόρτς, ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Ήθελα να σας προειδοποιήσω για το αυτή η προσπάθεια που κάνετε να παρουσιάσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για μια ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η οποία έχει παραστάτη και προστάτη ανθρώπους όπως τον κύριο Φερχόφστατ δεν συμβαίνει αυτό και δεν φοβόμαστε εμείς που ζούμε. Και επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη σεβασμού προς την βούληση των ε, Βρετανών που έχει ήδη εκφραστεί και η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή, τότε τρομάζουμε. Γι' αυτό ήθελα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει προσπάθεια καλής θέλησης από όλους γιατί θα πρέπει να συμβιώσουμε με τους Βρετανούς οι οποίοι είναι σημαντικό κομμάτι της άμυνας στο δυτικό κόσμο, του δυτικού κόσμου και με αυτούς θα πρέπει να μοιραστούμε ακόμα πολλά. Όχι μόνο εμπόριο και αγορές, όχι μόνο άμυνα, αλλά και το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ, έχει λήξει ο χρόνος σας. for minute. Εκτός μικροφώνου, ο επόμενος ομιλητής. Do you want to say something to me? Εκτός μικροφώνου ο ομιλητής. Sorry, colleagues, please. Συνάδελφοι, λέει η πρόεδρος, δεν είστε στον κατάλογο ομιλητών. Αν είχατε ζητήσει όμως, θα σας είχα δώσει το λόγο. Θα συνεχίσω λοιπόν για να μην ε, μείνουμε χωρίς χρόνο. Επόμενος ομιλητής, κύριος Κόσμο, για ένα λεπτό. Οι Βρετανοί ήδη εκφράστηκαν ε, στη διάρκεια ενός δημοψηφίσματος και για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να τους πιέζει ούτε να προσπαθεί να τους αλλάξει ε, την άποψη εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα. Είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί αυτό σημαίνει σεβασμό στη δημοκρατία. Και οποιαδήποτε παρέμβαση δεν συμφωνεί με αυτό δεν αποτελούν θετική εισφορά στο να καταλήξουμε σε μια φιλική ε, λύση που θα διαπραγματευτούμε για τον Brexit. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, παρακολουθήσει την ανευθυνότητα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου που θέλει μία άτακτη ε, έξοδο και αποχώρηση που θα διακυβεύσει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και που αμφισβητεί τα δικαιώματα των Ευρωπαίων ε, πολιτών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως επίσης και των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν, ξεκινώντας από εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπερασπιστούμε τους πολίτες αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιγιάν Μον, για ένα λεπτό. Αναφερθήκατε στη σημασία του να δούμε τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει το Brexit για τις δύο πλευρές, σε πολλούς κλάδους. Εγώ θα μιλήσω για τις αλληλευτικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο καλά γνωρίζει ο κύριος Μπαρνιέ, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Αν λοιπόν τεθεί σε εφαρμογή η η συμφωνία απαχώρησης και η μεταβατική, θα πρέπει να μειώσουμε τις συνέπειες για το στόλο μας που αλλιεύει στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για όλους, για να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε πρόσβαση στα ύδατα αυτά, τουλάχιστον με προσωρινικό τρόπο, μέχρι να διαπραγματευτούμε τη σχέση μας για το μέλλον. Ξέρω πως δεν σας αρέσει αυτό, αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε. Εδώ θα σταθώ για ένα λεπτό και θα πω πως πρέπει να τονίσω πως ένας από τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να έχουμε μια συμφωνία που θα επιτρέψει την αμοιβαία πρόσβαση σε ύδατα και αλληλευτικούς πόρους. Η συμφωνία αυτή έχει επίσης το πλεονέκτημα για όλους τους αλλοίς και θα επέτρεπε, λυπάμαι, πρέπει να σταματήσετε γιατί τελείωσε ο χρόνος σας. Ο κύριος Βουέλς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η υπεράσπιση κάθε χώρας και η άμυνα κάθε χώρας είναι χαρακτηριστικό της κυριαρχίας της χώρας αυτής και θεμελιώδης ευθύνη της κυβέρνησής της. Η κυβέρνηση ΜΕΙ συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το δημοψήφισμα και αυτό στην ουσία παρέδωσε τις ικανότητες, τις αμυντικές και τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών της χώρα σε ανεξέλεγκτους επιτρόπους. Είναι σαφές αυτό και στις ρήτρε 104 με 106 που περιλαμβάνονται στο 184 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Ανησυχώ γιατί και οι Βρετανοί συνάδελφοι απέτυχαν να κατανοήσουν την απειλή αυτή και γι' αυτό ζητώ από τους ε, συναδέλφους στο Westminster να απορρίψουν κάθε δυνατότητα επιστροφής στην απέσια αυτή συμφωνία. Η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα είδαμε να κρύβεται στο Λουξεμβούργο ο Βρετανός Πρωθυπουργό. Κρύβεται από την κοινοβουλευτική συζήτηση, κρύβεται από το κοινοβούλιο του. Κατά τα άλλα η δημοκρατία εδώ λειτουργεί και εκφράζονται οι απόψεις και με τις οποίες συμφωνούμε και με τις οποίες διαφωνούμε. Από το 2016 είχαμε πετύχει ε, μια καλή συμφωνία για μια ξεκάθαρη αποχώρηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη αποχώρηση. Η αποχώρηση κάτω από τις συνθήκες αυτές από την βορειοανατολική Αγγλία μέχρι το Φόκλαντς θα επηρεαστούν αρνητικά από την συμφωνία αυτή, την έλλειψή της περισσότερο. Αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα πράγματα από βρετανικής πλευράς δεν έχουν την εντολή πια να το κάνουν και ο βετανικός λαός πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Ε, τελείωσε η διαδικασία του Catch και γι' αυτό δίνουμε το λόγο για την απάντησή του στον βασικό διαπραγματευτή τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να είμαι σύντομος, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά πρέπει και να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος του Πρόεδρου Γιούνκερ και εξ ονόματος της διαπραγματευτικής ομάδας της, της, της οποίας είμαι υπεύθυνος τους τελευταίους, τα τελευταία τρία χρόνια. Φυσικά κατανοώ να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τέτοιες συζητήσεις είναι στιγμές αλήθειας. Τρία χρόνια μετά από το Brexit, από, την, το δημοψήφισμα, βρισκόμαστε σε μια στιγμή κρίσιμη. Πρέπει να είμαστε γαλήνοι και να σεβόμαστε οι μεν τους δε. Ε, εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά όσους πήραν το λόγο. Άκουσα ειδικά ε, τους ε, Ιρλανδούς και Βόρειο Ιρλανδούς ε, κοινοβουλευτικούς που είναι η πιο επικίνδυνη αν θέλετε κατάσταση που μπορεί να προκληθεί λόγω του Brexit. Άκουσα αυτά που είπατε για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άκουσα αυτά τα οποία είπαμε για την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς και τις τέσσερις ελευθερίες που τη συνοδεύουν. Άκουσα επίσης προσεκτικά και αυτούς οι οποίοι είχαν διαφορετική άποψη. Και υπάρχει μια κατηγορία στην οποία, η οποία μου απευθύνθηκε και πρέπει να απαντήσω. Και το λέω στον κύριο Τσάνι που δεν είναι εδώ, στον κύριο Φάρατ, στον κύριο Μάντισον και σε άλλους. Κανείς, μα κανείς δεν θέλει να αγνοήσει την επιλογή της πλειοψηφίας ε, του Βρετανικού λαού. Κανένας δεν θέλει να αλλάξει το Brexit. Κανένας δεν θέλει να διατηρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την θέλησή του, στην Τελωνιακή Ένωση ή στην εσωτερική αγορά. Είναι η δική σας ευθύνη ε, που πήρατε και θέλετε να φύγετε, λυπούμεθα γι' αυτό και το λέμε πάντα εγώ ποτέ δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτή τη κίνησή σας, αλλά το σεβόμαστε. Η εντολή την οποία πάντα είχα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από το Κοινοβούλιο και η εντολή την οποία ασκώ αν θέλετε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βρούμε μία συμφωνία. Αυτό απαιτεί δύο πράγματα κυρίες και κύριοι. Πρώτον να πούμε την αλήθεια εδώ στο Κοινοβούλιο, στους πολίτες για τις συνέπειες του Brexit. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αναφερθήκατε στον σεβασμό των βετανών πολιτών, όπως και άλλων, όλων των πολιτών, έχουν δικαίωμα στην αλήθεια, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις συνέπειες ε, του Brexit που είναι πολύ πιο σοβαρές από αυτές τις οποίες του έχετε πει μέχρι τώρα του πολίτη. Τι θα ακολουθήσει μετά από το Brexit. Θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και εμείς επίσης. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τις συνέπειες του Brexit με συμφωνία την οποία επιθυμούμε και για την οποία εργαζόμαστε και τις συνέπειες ε, του Brexit χωρίς συμφωνία. Να πω στον κύριο Νιούτον Τάν, όπως και σε άλλους, ότι έχουμε προετοιμαστεί για την υπόθεση του Brexit χωρίς συμφωνία και στον τομέα της συνεργασίας ε, της Europol. Φυσικά το no deal δεν είναι μια τελική αν θέλετε κατάληξη, είναι μια προσωρινή λύση έτσι ώστε να βρεθεί ε, ε, κάποια συμφωνία. Αυτό κάνω εδώ και τρία χρόνια, να λέω την αλήθεια, να λέω την αλήθεια σε όλους. Και η αλήθεια έχει απαιτήσει. Απαιτεί να βρεθούν νομικές λύσεις, γιατί κάνουμε μια συνθήκη, δεν κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, δεν κάνουμε μια διακήρυξη. Θέλουμε να βρούμε σοβαρές νομικές λύσεις στα θέματα τα οποία τίθενται λόγω του διαζυγίου που εσείς επιλέξατε, λόγω του Brexit λύσεις και στην Ιρλανδία και σε άλλους τομείς όπως η αλία. Πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες να είναι συγκεκριμένες, να είναι λειτουργικές και να μην είναι ε, θα έλεγα απλές γενικόλογες δηλώσεις. Αυτό περιμένουμε και από τον Πρωθυπουργό Τζόνσον και την ομάδα του. Αν αμφισβητείτε το backstop ή μια κάποια άλλη ρύθμιση, δώστε τις προτάσεις σας, δώστε τις απαντήσεις σας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κανένας δεν θα πρέπει να αμφισβητήσει την διαθεσιμότητά μας και όσο μας έχετε εμπιστοσύνη εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε ε, διάθεση και με κάθε ειλικρίνεια. Ευχαριστώ τον Μισελ Μπαρνιέ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Τούπερα, η ενεκπρόσωπο του Συμβουλίου. Έχετε τον λόγο. Mr. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, παρόλα Παρόλη την αβεβαιότητα από την πλευρά του Εμένου Βασιλείου, εμεί θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, εάν αυτές μας οδηγήσουν στο ε, να βρούμε μια λύση η οποία θα συμμορφώνεται με τις αρχές μας. Μια συντεταγμένη αποχώρηση του Ευρωπαϊκού, του με του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την προτεραιότητά μας μέχρι την τελευταία στιγμή δεδομένων των αρνητικών συνεπειών ενός σκληρού Brexit και μέχρι τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα στοχευμένα μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσουμε την ενδεχόμενη, ε, τις ενδεχόμενες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και την παράταση της ε, προθεσμίας για το άρθρο 50 εάν λάβουμε μία ε, αιτιολογημένη, ε, ένα αιτιολογημένο αίτημα από τη Βρετανική κυβέρνηση. Να σας υπενθυμίσω πως η υπομονή αποτελεί αρετή. Βασιζόμαστε στη δική σας συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ για τις απόψεις σας, για τα σχόλιά σας και για την προσοχή με την οποία μας ακούσατε κυρίες και κύριοι. Grazie. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω δύο προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή. Η συζήτηση περατώνεται εδώ λοιπόν και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ένα λεπτό διακοπή όμως προηγουμένως, ώστε να μπουν οι συνάδελφοι και να καθίσουν. Ένα λεπτό διακοπή. Allora riprendiamo. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία και η μία γεγραμμένη ανακοίνωσαν αποφάσεις για αλλαγές στους ορισμούς σε διάφορες αντιπροσωπείες. Οι αποφάσεις αυτές επισυνάπτονται στα σημερινά πρακτικά και θα αρχίσουν να ισχύουν από τώρα από τη στιγμή της ανακοίνωσης δηλαδή. Τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στις ψηφοφορίες. Έκθεση Howard, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Τροπολογία αριθμός 1, μία ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Hanno votato tutti. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της προφορίας. Εγκρίνεται. Πάλι έκθεση Howard, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού ε, το λόγο ο εισηγητής παρακαλώ. Δύο λεπτά. Παρακαλώ. Δεν είναι εδώ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις εισηγητές και τη γραμματεία για τη δουλειά που έχουν βάλει σε αυτή την έκθεση και θέλω να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Ο τροποποιημένο αυτό αριθμό 2 προπολογισμό είναι κάπω διαφορετικό από του συνηθισμένου. και ε, έχει επηρεαστεί και από το ε, συμπληρωματικό προπολογισμό του 2019 μετά από διαβουλεύσει των χωρών μελών ε, με το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Θα υπάρξει λοιπόν αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2019, αριθμός 2, για να καλυφθούν δύο προγράμματα ώστε να λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, οικονομία και το Έρασμος ε, και το 2020 που είναι δύο προγράμματα τα οποία αποτελούν την προστιθέμενη αξία με 20 εκατομμύρια το πρώτο και 8 το δεύτερο παραπάνω. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και άλλα θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Ο προπολογισμό αυτός αντικατοπτρίζει την αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε μαζί πολύ περισσότερα από ότι κάθε μία χωριστά χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να πετύχει. Ζητώ τη στήριξή σα λοιπόν. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει ονομαστικά. Άρχεται. Ψηφίσετε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μούρεσεν για την κινητοποίηση του Ταμείου Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαία ψηφοφορία, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Χάουαρτ. ξανά σχέδιο διευθυντικού προϋπολογισμού 3. Μία ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ζόγκα. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Μία ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματο για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγραφος 4. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα Διαναστα... των χειρών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο, τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήματα. Διανατάσσεως των χειρών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 παράγραφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη δέλτα, δύο τμήματα. Πρώτη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη κάπα, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη εν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη πληροφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Περιμένουμε τις αιτιολογήσεις ε, ψήφου. Διακόπτεται για λίγα λεπτά η συνεδρίαση. Ευχαριστώ. όλα σεδούτα. ξαναρχίζουμε τη συνεδρίαση για τι δηλώσει ψήφου, για τι ανακοινώσει ψήφου. Οι συνάδελφοι που δεν θέλουν να μετάσχουν παρακαλώ να βγουν έξω για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά η συνεδρίαση τη ολομέλεια. Συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε με τι αιτιολογήσει ψήφου. Take part to the operation to leave the plenary. Βγείτε από την αίθουσα παρακαλώ όσοι δεν θέλετε να συμμετάσχετε στις συζητήσεις. Αυτό είναι θέμα αυροφροσύνης προς την συναδέλφους σας. Dear colleagues, I kindly ask you again to leave the plenary if you are not... Βγείτε από την αίθουσα παρακαλώ αν δεν θέλετε να μετάσχετε στη διαδικασία αιτιολόγησης ψήφου. Procediamo con le dichiarazioni di Συνεχίζουμε <clears throat> με τις ε, αιτιολογήσεις ψήφου. Για την πρόταση ψηφίσματος για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τεντάρλινγκ, ένα λεπτό. Δεν θέλει να μιλήσει η συνάδελφος Κίρτεν Ντάμεν. Συνεχίζουμε. Φώναρα. Ένα λεπτό. It does not work. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Λειτουργεί. Ευχαριστώ. Για το ψήφισμα για τη Βρετανία ψήφισα ξανά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας τη μελλοντική μας σχέση με την Βρετανία. Να μην υπάρχει σύγκρουση. Να επιβάλλουμε, δεν πρέπει να επιβάλλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να υιοθετήσει μια συμφωνία που τρεις φορές απέριψε. Θυμάμαι στην Τσεχοσλοβακία είχαμε μια, ένα επιτυχές διαζύγιο μεταξύ Τσεχίας και Σλοβακίας. Για να έχει ένα καλό διαζύγιο πρέπει να υπάρχει μια γενεοδορία από τις δύο πλευρές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ. Αλλιώ, χωρίς τη γενεοδορία της Ευρώπης, το, το διαζύγιο θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ ε, προβληματικό. Ευχαριστώ. Σόντροβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Από την ίδια χώρα με τον συνάδελφο Βόντρα ε, προέρχομαι, αλλά εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα ακριβώ γιατί σέβομαι το ψήφισμα του Βρετανικού Κοινοβουλίου που λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να εγκαταλείψει την Ένωση χωρί συμφωνία. Αυτό είναι ο λόγο πιστεύω για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε σωστά με την πρότασή του για μια καθυστέρηση σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Εμείς δεν επιβάλλουμε κάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν επιβάλλουμε τη δική μας συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που υπέγραψε και η Βρετανή Πρωθυπουργός το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να υποβάλει τροπολογίε στην συμφωνία αυτή, μπορεί να κάνει αλλαγές. Ο Πρωθυπουργό, ωστόσο, τη Βρετανία δεν έχει προτείνει αλλαγέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει μεγάλη υπομονή, όπω και ο διαπραγματευτή Μπαρνιέ, για να υπάρξει μια τελική συμφωνία, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο έρθει με συγκεκριμένε προτάσει αλλαγή. Ευχαριστώ. Πόριτ, ένα λεπτό. microphone's not coming on. I have. Now it's working. It's not coming on. Okay. I have voted. Στηρίζω το ψήφισμα, όχι γιατί θέλω να υλοποιηθεί η συμφωνία αποχώρησης, γιατί οποιαδήποτε μορφή Brexit είναι ζημιογόνος για όλου. Αλλά επειδή το κείμενο ε, δεν αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξει παράταση προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία και να ολοκληρωθεί αυτή η δημοκρατική διαδικασία με νέο δημοψήφισμα ή με νέες εκλογές ή με την ανάκληση του άρθρου 50. Όλοι οι Ευρωπαίοι λοιπόν εδώ πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν την αλληλεγγύη τους απέναντί μας και να μην υπάρχει πια αυτός ο κίνδυνος ο λαϊκίστικος εκεί από τα δεξιά του σώματος που το μόνο που κάνουν εδώ είναι ότι πατάνε για να παίρνουν τα επιδόματά τους και τις αποζημιώσεις τους. Πρέπει να σκεφτούμε το εθνικό συμφέρον. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό από τον αριθμό 10 της Downing Street, από την κατοικία του Πρωθυπουργού όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σαν αποτέλεσμα την ομοιρία όλων μας. Όπως είπανε και συνάδελφοι που έχουμε εδώ την πλειοψηφία, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αποφύγουμε τον αθλητισμό και τον λαϊκισμό και να μην τον αφήσουμε να νικήσει. Συνάδελφοι, παρακαλώ να σέβεστε το ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πάτεν, ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου, κύριος Πάτεν. Καταψήφισα ε, κατά αυτήν την αυτό το, το, το, κατολικό ψήφισμα του κυρίου Βερχόφστα. Θεωρώ δηλαδή πως θα πρέπει να έχουμε ένα καθαρό Brexit. Και αυτό γιατί, γιατί το 58% των ε, Midlands ε, ε, υποστήριξε κάτι τέτοιο και αντίστοιχα ποσοστά είχαμε και σε άλλες περιοχές. το, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ποσοστό η δημοκρατική πλειοψηφία της χώρας μου υπερψήφισε το να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άκουσα τώρα κατά τις τελευταίες τρεις ώρες διάφορους ευρωβουλευτές να αναφέρουν και να λένε ότι αυτό ο λαό δεν ξέρει τι κάνει και ότι θα πρέπει να ακούσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο όταν συμφωνεί με αυτό εδώ το θεσμικό όργανο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε μόνο μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχει δημοκρατία. Ο κύριος Μπαρνιέ είπε και το κατέστησε σαφέ ότι οποιοδήποτε και αν είναι το backstop, αν εφαρμοστεί ή όχι, δεν υπάρχει ε, καμία, κανένας τρόπος να ξεφύγουν από την Τελωνιακή Ένωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα 17,4 εκατομμύρια των Βρετανών που ψήφισαν την αποχώρηση από τον Brexit. Έφτασε όμως η ώρα να γίνει αυτό το καθαρό Brexit και να αποχωρήσουμε επιτέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Χουκ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, στήριξα το ψήφισμα σήμερα γιατί αναγνωρίζει τις ε, προοπτικές ανάκλησης του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί δεν έχει πλειοψηφία ο Μπόρις ε, Τζόνσον στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, γι' αυτό και θέλησε να το κλείσει και γι' αυτό θέλει να εμποδίσει τον κόσμο να ψηφίσει για μια συγκεκριμένη συμφωνία αποχώρησης το δημοψήφισμα του 2016 δεν ήταν ξεκάθαρο και πάρα πολλά ψέματα και παραπληροφόρηση υπήρχε. Για παράδειγμα, ότι θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα Τούρκου ευρωβουλευτέ. Ο Τζόνσον είπε ότι ήταν εύκολο να αποχωρήσουν. Ε, αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Η απόφαση του 2016 είναι παλιά, παροχημένη και το 2019 είμαστε διαφορετικοί. Κανείς από τους νέους δεν θέλει να μειωθούν οι δαπάνες ε, στην ιατρική κάλυψη, για παράδειγμα, όπως τελικά κάνει η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε μια μεγάλη χώρα και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βάλουμε πίσω το Brexit, να γίνει παρελθόν και να μην ισχύσει. Μπέρντερ, ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σήμερα υπερψήφισα το ψήφισμα ε, για το, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ δεν θέλω τον Brexit, το μισό. Οποιαδήποτε συμφωνία όμως πρέπει να περάσει από τον κόσμο. Ο Μπόρις Τζόνσον ε, παίζει παιχνίδια ε, προς όφελος δικό του και μόνο. Ο κόσμος θέλει να σταματήσει αυτή η διαδικασία Μπρίξον και εγώ και οι σοσιαλδημοκράτες ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες, αγαπάμε τους Ευρωπαίους πολίτες και θέλουμε να ανακληθεί το άρθρο 5 και να σταματήσει το Brexit και αυτή η διαδικασία. Θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ψήφισμα αναγνωρίζει την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους Βρετανούς, οι οποίοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, αλλά η αναταραχή είναι τεράστια. Τώρα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Εγώ και όλοι εμείς θα είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ευχαρίστως να φροντίσουμε να ανακληθεί το άρθρο 50 και να είμαστε πλήρως μέλη εδώ. Γκίμψεν για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο, κύριε Γκίμψεν. Ευχαριστώ. Υποστήριξα το ψήφισμα και ζήτησα την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υποστηρίζω καμία συμφωνία για το Brexit με ή Χωρί συμφωνία. Κάθε Brexit είναι κακό και για τη Βρετανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσω να κάνω καμπάνια για να σταματήσει το Brexit. Αυτή αυτό το ψήφισμα όμως είναι σημαντικό γιατί αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο για να επιβάλλει στην κυβέρνηση να ζητήσει παράταση σε περίπτωση ε, εξόδου χωρίς συμφωνία. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν δρά υπέρ των Ευρωπαίων των πολιτών της Βρετανίας, έκλεισε το κοινοβούλιο, δηλώνει ότι θα παραβιάσει τον νόμο σε περίπτωση που δεν, που δεν υπάρξει ε, συμφωνία, δρά ως δικτάτορας είναι καιρός να τον ρίξουμε μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Ευχαριστώ. Χάουερθ, ένα λεπτό. Δεν ήταν αυτό το πλάνο. Αντί από πραγματικά προγράμματα αποχωρήσει το μόνο το καλύτερο που μας παρέχουν είναι η επιβίωση. Βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης σε εξαιρετικά αδύναμη θέση ή και καμία συμφωνία. Λέγανε ότι θα έχουμε την κυριαρχία μας και βλέπουμε την ε, ισχύ που έχει ένας ισχυρός γείτονας που επιβάλλει, ε, που επιβάλλει αυτό που θεωρεί και εμείς λίγα μπορούμε να κάνουμε χάνονται θέσεις στη βιομηχανία. Τα δικαιώματα των πολιτών κάθε πολίτη της Ευρώπης μειώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα του Brexit. Καθόλου αυτά που έλεγαν πριν το δημοψήφισμα και με το οποίο κέρδισαν το δημοψήφισμα. Έξω από την Ένωση θα καταλάβουμε πολύ γρήγορα ότι τους περιορισμούς της εθνικής κυριαρχίας έξω από την Ευρώπη. Ακούμε πολλά για τη δημοκρατία, αλλά τι γίνεται με τη λογοδοσία. Τι συμβαίνει με αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τις, υποσχέσει τις υποσχέσεις τους. Ας ξαναπαρουσιάσουμε στο Βρετανικό λαό την πραγματικότητα και θα του ζητήσουμε να αποφασίσει με βάση την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Χίβερ, ένα λεπτό. Μετά από όλα αυτά τα παράξενα και τα περίεργα που ακούσαμε, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους πως ο κύριος Φαράζ εκπροσωπεί το μεγάλο κομμάτι εκείνων που είναι υπέρ του Brexit στη χώρα μου. Σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση ψηφίσματο, ε, πραγματικά εσεί λέτε ότι είναι κάτι το δυσάρεστο ε, το ότι κάνουμε αυτό το Brexit, αλλά αυτή είναι η δική σα άποψη. Εκείνοι που υποστηρίζουν το Brexit, οι Βρετανοί ε, πολίτε, δεν έχουν την ίδια άποψη. Βλέπετε λοιπόν ε, εμείς που είμαστε οι Brexiters, που είμαστε δηλαδή υπέρ του Brexit ε, κάνουμε τη φωνή μας ακουστή και εκπροσωπούμε την, τους, την Βρετανική πλειοψηφία δηλαδή ε, ακούσαμε το τι λέτε και πραγματικά είναι αστεία τα όσα λέτε. Το κόμμα του Brexit έχει ε, ταχθεί ιστορικά υπέρ τη εξόδου και τώρα αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα καθαρό Brexit και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή η υποστήριξη για το να μην υπάρξει συμφωνία και έξοδος με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται όλο και περισσότερο και πραγματικά θα, αυτή τη φορά θα καταφέρουμε και θα αποχωρήσουμε πράγματι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ ένα λεπτό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτό το εξαιρετικό δημοκρατικό θεσμικό όργανο που υποστηρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζει μια περαιτέρω παράταση τη εφαρμογή του άρθρου 50. Μια συμφωνία δηλαδή, μια μάλλον έξοδο ε, Brexit χωρί ε, συμφωνία θα ήταν ε, τραγική, ειδικότερα για τι πιο ευάλωτε ομάδε πολιτών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά του πολίτε εκείνου οι οποίοι εξαρτώνται από την εισαγωγή φαρμακευτικών συμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ζωέ δηλαδή πολλών ανθρώπων εξαρτώνται από την εύρυθμη και σωστή εισαγωγή φαρμακευτικών συμβασμάτων αποτέλεσμα Κανένα δεν μπορεί λοιπόν να εγγυηθεί ότι αυτά τα φάρμακα θα είναι δυνατό να ε, συνεχίσουν να εισέρχονται ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αν δεν υπάρξει συμφωνία ε, μέσα στο Brexit. Και πραγματικά το να θέλει κανεί να θέσει τα δικά του συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα αυτών των ευάλωτων ε, πολιτών είναι κάτι το ε, σοκαριστικό και νομίζω πως έχει οδηγήσει πολλούς εδώ ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιταχθούν σε ένα τέτοιο Brexit χωρίς συμφωνία. Κανένας δεν υποστήριξε κάτι τέτοιο και κανένας δεν υποστήριξε το να αρνηθούμε την παροχή κρίσιμων φαρμάκων στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας. δηλαδή μία έξοδος χωρίς συμφωνία θα αποτελέσει μια κακή συμφωνία, ένα κακό για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ντόγνε για ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τι ωραία που βλέπω ότι είναι εδώ οι Βρετανοί και μπήκανε πριν για να ψεφίσουν πριν στη συζήτηση που ήτανε. Κατά τα άλλα, ψέματα, λάθη, μισές αλήθειες, κατηγορίες, υποθέσεις ότι η Βρετανία βρίσκεται υπό δικτατορία. Μα οι δικτάτορες δεν προσφέρουν εκλογές, δεν λένε να γίνουν εκλογές και όταν λένε να γίνουν εκλογές εσείς δεν τις δεχκέστε, λέτε όχι να μην γίνουνε. Γιατί ξέρετε ότι θα χάσετε. Κύριο Στάσφελτ, εκεί που είμαι εγώ και που έχει καταστραφεί ο κύριο Κόρμπιν, το 70% του κόσμου στο Άσφιλ ψήφισαν Brexit, να αποχωρήσουμε. Αλλά δεν ενδιαφέρεται εδώ το σώμα για τη φωνή των Βρετανών, για το τι ψήφισαν. Δεν ε, προσωπούνται εδώ οι Βρετανοί και η φωνή τους. Φεύγουμε. Ο and bye, ο Ρεβουάρ. Ευχαριστώ. Πάλμερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Την Πρόεδρε θα τα πω τα πράγματα ως έχουν. Γιατί η διατύπωση του ψηφίσματος αυτού είναι στενή. Για το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών και την προστασία των, Ευρωπαίων πολιτών στον Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεταχείριση των ανθρώπων αυτών είναι ιδιαίτερα ατυχής και πραγματικά ντρέπομαι για τη χώρα μου γι' αυτό, για τη χώρα που αγαπάω για τη χώρα που αγαπούν εξίσου όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που την έκαναν ε, ε, δικιά τους χώρα, που πληρώνουν φόρους, που ζουν, εργάζονται, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό το σχέδιο που προβλέπετε. Για όλους αυτούς λοιπόν τους Ευρωπαίους στον Ενωμένο Βασίλειο που εκπροσωπώ στα Midland, Θέλω να πω ότι η χώρα μου είναι κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε και σίγουρα όλοι αυτοί οι πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν τώρα. Ο κύριος η κυρία Μπρόφη για ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, υπερψήφισε το ψήφισμα. Δεν θέλω ωστόσο να υπάρξει Brexit. Για δύο δεκαετίες ήμουν επαγγελματία στην Βρετανία και το βασικό θέμα που έβλεπα ότι ήταν θετικό ήταν τα κοινωνικά δικαιώματα και τα ζητήματα απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν επαγγελματία στον τομέα της υγείας βλέπω τους κινδύνους του εθνικού συστήματος υγείας λόγω του Brexit. 5,5% ε, μείωση έχει τα τελευταία χρόνια και αυτό θα μειωθεί και ο αριθμό των εργαζομένων στον τομέα τη υγεία θα μειωθεί σημαντικά εάν αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περισσότερο αν δεν υπάρξει συμφωνία. Είναι ευπρόσδεκτη η συμφωνία αυτή. Θα δώσει διαβεβαιώσει στου Ευρωπαίου πολίτε που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία αλλά η, αποχω... η μη αποχώρηση θα πρέπει να μείνει η πρώτη προτεραιότητά μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Bonding, ένα λεπτό. Έχει το λόγο. Λειτουργεί, έτσι. Συνάδελφοι, αυτή ήταν η πιο δύσκολη ψηφοφορία που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Υποστηρίζω απόλυτα τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για μια παράταση του άρθρου 50 αλλά κάθε συμφωνία αποχώρησης πρέπει να επανέλθει στους πολίτες της, Ένωσης, της Βρετανίας στο, σε ένα δημοψήφισμα που θα έχει και την επιλογή της παραμονής στην Ένωση. Μόνο με αυτό, και είμαι, είμαι βέβαιη ότι αυτή τη, φορά θα κερδίσουμε, γιατί αυτή σήμερα οι νέοι θα έρθουν να ψηφίσουν. Είναι οργισμένοι αυτή τη στιγμή. Τα τρία τέταρτα από αυτούς ήταν πολύ νέοι, δεν είχαν ψηφίσει το 2015 το 2016. Ε, τώρα έφτασαν στην ηλικία ενηλικίωσης και κατά τα τρία τέταρτα υποστηρίζουν την παραμονή της Βρετανίας στην Ένωση. Παρακαλώ συνάδελφοι, επιστρέψτε στις πατρίδες σας και πιέστε τους ηγέτες σας να δώσουν στους Βρετανούς πολίτες μια ευκαιρία να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μπάνιεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί υποστήριξα μια πρόταση ψηφίσματος ε, που ε, υποστηρίζει ουσιαστικά το αποτέλεσμα μια συμφωνία η οποία έτυχε διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κόλλησε εντό εισαγωγικών στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι, λοιπόν, ο λόγο είναι ότι δίνει λοιπόν τη δυνατότητα ε, στο, Ευρωπαϊκό, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει τη δική του άποψη, καθώ παρέχει ακριβώ μια παράταση τη εφαρμογή του άρθρου 50, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει τη δική του θέση. μια έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί συμφωνία θα μπορούσε μπορούσε αποτελέσει καταστροφή για τον αγροτικό μα ε, τομέα. Δηλαδή, το 97% των εξαγωγών των αγροτικών μα ε, προϊόντων κατευθύνεται προ τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση ε, εξάγουμε βόλιο κρέα, δημητριακά και πολλά άλλα τρόφιμα. Οπότε το να χάσουμε την πρόσβαση σε αυτέ τι αγορέ δεν θα ήταν προ το καλύτερο συμφέρον των πολιτών μου. Και γι' αυτό θεωρώ πω η προτεραιότητα αποτελεί το να μην υποστηρίξουμε μια έξοδο χωρί συμφωνία. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ιδιότητα του μέλου του Ηνωμένου Βασιλείου της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντέιβις, για ένα λεπτό. Κύριε Ντέιβις, έχετε το λόγο. To... Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να διαχειριστούμε το ε, Brexit, θέλω να σταματήσουμε το Brexit. Εδώ, σε αυτό το θεσμικό όργανο, υποστηρίζουμε τι ε, δημοκρατικέ αξίε, αλλά εγώ υποστηρίζω και τι φιλελεύθερε αξίε. Δηλαδή, υποστηρίζουμε μια οικονομία η οποία αποβαίνει προ όφελο όλων και είμαστε υπέρ μέτρων που προστατεύουν του πάντε. Δεν θέλω λοιπόν η δική μου χώρα να αποκλειστεί από. Ε, τι αίθουσε στι οποίε θα λαμβάνονται οι πιο σημαντικέ αποφάσει για αυτά τα ζητήματα και δεν θέλω να φύγουμε τρέχοντα από τη λήψη αυτών των σημαντικών αποφάσεων. Θέλω να παραμείνουμε στην καρδιά ε, τη χάραξη τη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να παραμείνουμε σε ηγετικό ρόλο. Οπότε είναι πολύ ξεκάθαρη δική μου θέση. Σε καμία περίπτωση Brexit. Adesso... Adesso la parola... Ευχαριστώ. Άντζου Σελίμπα. Για ένα λεπτό. Το Brexit ως ε, σπάθα πάνω από το κεφάλι μας αποτελεί απειλή για όλους μας. Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα είναι μια καταστροφή που πρέπει να αποφύγουμε. Δυστυχώς οι αβεβαιότητες, ε, η πολιτική αστάθεια αυξάνεται κάθε στιγμή. Με αυτή την κατάσταση πώς θα διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και τις επιλογές των ε, Βρετανών ε, πολιτών που ζουν ε, στην υπόλοιπη Ευρώπη, των Ευρωπαίων που ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Επίση, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα κάνει μεγάλη ζημιά στι επιχειρήσει, στην απασχόληση τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη προτεραιότητά μα είναι να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει και του εργαζόμενου, ώστε το κόστο και ε, τα βάρη και ζημιά να περιοριστούν στο ελάχιστο. Επίσης, ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες στα σύνορα εκεί. Ε, πρέπει και αυτές να περιοριστούν στο ελάχιστο. Γι' αυτό χρειάζεται επικοδομητικός διάλογος για να αποφύγουμε την αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Και αυτό πρέπει να βρίσκεται ε, κατά προτεραιότητα πάνω από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε. Νταμίζα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ο κύριος Ταμίζα. Ευχαριστώ. Ω επιχειρηματία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οποιοδήποτε επιχειρηματίας θα ήθελε να χάσει μια αγορά 515 εκατομμυρίων για 65 εκατομμύρια αγορά. Είναι τεράστια διαφορά. Εγώ έχω φτιάξει την ύποκος.com και σε πέντε χρόνια έγινε μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων. Και ο λόγος είναι γιατί είχαμε μια αγορά 300 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλιώς θα πουλάμε σε 60 εκατομμύρια. Τότε δεν θα τα είχαμε καταφέρει το ίδιο. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες λοιπόν τώρα, αν υπάρξει το Brexit, είναι ότι θα φτιάξουν ένα γραφείο στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, στο Δουβλίνο και η απασχόληση θα φύγει και θα πάει σε αυτές τις πόλεις. Δηλαδή πυροβολούμε τον εαυτό μας στα πόδια. Σκάβουμε το λάκκο μας. Βόντεν, ένα λεπτό. Ο κύριος Πάτον προφανώς δεν καταλαβαίνει το 62% των ψηφοφόρων δεν σημαίνει 62% του κόσμου. Ψέματα, όπως πάντα. Όπως είδαμε και στο σκάνδαλο Windows, η κυβέρνησή μας ε, κάνει ό,τι μπορεί να χωρίζει τις οικογένειες και αυτό προτίθεται να κάνει και τώρα. Η Ευρώπη είναι μια οικογένεια εθνών και λαών που αν επιτρέψουμε στους τόροι να διαιρέσει την οικογένεια αυτή θα δημιουργήσει τεράστια βλάβη και σε εμά και στους Ευρωπαίους. Όπως το Brexit θα διαιρέσει την ευρωπαϊκή οικογένεια, ταυτόχρονα θα διαιρέσει και την Βρετανία. Εγώ είμαι Βρετανή γεννημένη στη Σκωτία. Αισθάνομαι παιδί δύο εθνοτήτων. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ηλικία 218 ε, έτη και ο κύριος Τζόνσον θέλει να υπονομεύσει αυτή την ένωση μαζί με, αγνοώντας ε, τις, φε, τα συμφέροντα της Βορείου Ιρλανδίας και αδιαφορώντας για τη Σκοτία. Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε ξανά μία, μία γενιά William Wallace να εμφανίζεται στη Σκοτία αν συνεχίσει ο Τζόνσον. Ρίτσι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. For this. 2 Είχα ψηφίσει τον, τον, ε, χτες προχτες, ε, ε, τον Ιούλιο θα γιορτάσει 20 χρόνια η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Το Σάββατο είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Μην ξεχνάτε ότι η συμφωνία αυτή ήταν η τελευταία συμφωνία ειρήνης, ειρήνευσης στην Ευρώπη και φοβάμαι ότι το Brexit θα οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις στην Βόρεια Ιρλανδία και προφανώς ο κύριος Φαράτζ δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Κέλλη για ένα λεπτό. Όχι διοθόνιο. Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω την ψηφοφορία η οποία μόλις τώρα έλαβε χώρα. Προφανώ ε, σέβομαι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο των Βρετανών πολιτών, αλλά από την άλλη ε, πλευρά ε, πραγματικά υποστηρίζω αυτό το ψήφισμα το οποίο θα επιτρέψει μια παράταση ε, της ε, προθεσμίας για το Brexit. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, και να σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου ότι δηλαδή το άρθρο 50 μπορεί να κληθεί μόνο μερός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποστηρίσουμε ε, τα δικαιώματα των όσων βιώνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, δεν θα πρέπει να αρνηθούμε ε, το δικαίωμα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζουν στις δύο πλευρές των συνόρων της Βορείου Ιρλανδίας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στα όσα λένε οι ευρωβουλευτές του κόμματος του Brexit, ότι δηλαδή ουσιαστικά ε, το ευρωπαϊκό σύστημα ψήφων τους επέτρεψε να έχουν αυτές τις έδρες που έχουν σήμερα. Με βάση το βρετανικό σύστημα δεν θα είχαν αυτές τις έδρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χάρηκα που συμμετείχα στη σημερινή συζήτηση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από τους ευρωβουλευτές εξήγησαν τις θέσεις τους, την άποψή τους για το backstop, ότι στηρίζουν τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και πόσο σημαντικό είναι να την προστατέψουμε. Στην ψηφοφορία 544 υπερψήφισαν αυτή τη συμφωνία που είναι μια μεγάλη πλειοψηφία στο σώμα. Χαίρομαι επίσης που ακούω ότι οι ευρωβουλευτές είναι διατεθειμένοι να δώσουν παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση που ο Μπόρις Τζόνσον το ζητήσει. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Χάναν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Οι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα, ίσως και χωρίς να το θέλουν, ε, μειώνουν τις πιθανότητες να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των υποχωρήσεων που δεν κάνουν, του μηχανισμού της ασύμετρης διαιτησίας. Το μόνο πράγμα που δεν θέλουν να δεχτούν εδώ πέρα οι ευρωβουλευτές είναι τον μηχανισμό αυτό αποχώρησης, γιατί επιμένουν στο backstop. Έτσι λοιπόν αυτή η δήλωση στο, στο, στο σώμα σήμερα έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες να επιτευχθεί κάποια συμφωνία αποχώρησης. Εδώ αυτή η κρίση για το Brexit, μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν έχουμε κρίση λόγω Brexit, έχουμε κρίση λόγω της άρνησης των ευρωβουλευτών που δεν θέλουν το Brexit να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Δεν θέλουν να κάνουν εκλογές. Ελπίζω τελικά να τα καταφέρουμε και να μην έχουμε παράπλευρες απώλειες. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Τόμτς. Πράγματι βρισκόμαστε πρώτων θυρών του Brexit, αλλά ε, τελικά ε, εκείνο που θα είναι το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ε, δεν θα υπάρχει κανένας ε, ε, ο οποίος θα κερδίσει από αυτά. Οπότε το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις ζημίες για όλους. Προφανώς και έχει νόημα να δοθεί μια περαιτέρω προθεσμία, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος για κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή λάβουν χώρα νέες εκλογές ή αν λάβει χώρα ένα νέο δημοψήφισμα. Το να δίνεται έτσι απλά η προθεσμία δεν ξέρω αν έχει νόημα. Πάντως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία το εξή για όλους μας. Ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις πολίτριες μας. Στην ε, ε, Ενωμένο ε, Βασίλειο ουσιαστικά παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποδιοπομπαίος τράγος που φταίει δηλαδή για, για όλα όσα συμβαίνουν. Ωστόσο, ουσιαστικά αν λάβει χώρα μία έξοδος χωρί συμφωνία, οι μόνοι οι οποίοι θα φταίνε γι' αυτό θα είναι η πολιτική του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. UK from Germany, Πρόεδρε, όταν πήγα πριν 20 χρόνια στη Βρετανία από την Γερμανία, έφτασα σε μια παγκοσμιοποιημένη Βρετανία που με καλωσόρισε με ανοιχτέ αγκαλιέ. Η συμμετοχή της Βρετανίας στην Ένωση μου επέτρεψε να χτίσω μια ζωή και να αποκτήσω ευκαιρίες σε μια χώρα που αγαπώ. Σήμερα όμως 3 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης στη Βρετανία αντιμετωπίζουν ένα κλίμα φόβου και αβεβαιότητας. Ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ότι δεν θα μειωθούν τα δικαιώματά τους από το Brexit, αλλά παρεύει αυτή την υπόσχεση όπως πολλές άλλες. Το πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης δεν είναι το ίδιο με τα δικαιώματα που έχουμε τώρα, δημιουργώντα πολλά προβλήματα, ιδίω ε, στους πιο ευάλωτους που δεν μπορούν εύκολα να αποδείξουν ότι μπορούν να υπαχθούν στο σύστημα αυτό. Πρέπει να έχουμε ένα εύκολο σύστημα με εύκολη καταχώρηση των ατόμων, όχι ένα σύστημα που κανείς πρέπει να βρει έγγραφα και έγγραφα πολλών ετών. Αλλιώς βρίσκουμε, ζούμε σε ένα νέο σκάνδαλο Windows σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γι' αυτό υπερψήφισα το ψήφισμα. Αλλά ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών στη Βρετανία είναι να σταματήσουμε τον Brexit. Ευχαριστώ. Thank you. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. αισθάνθηκα βλέποντας και ποιοι μιλάνε ότι είμαι σαν ε, αντιπρόεδρος στο, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Διακόπτουν τις συνεδρίες, ξαναρχίζουμε στις 3. Ευχαριστώ.

Ευχαριστώ,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 Good afternoon, colleagues. Χαίρετε. τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που ενεκρίθησαν είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν σχόλια για τα πρακτικά και τα κείμενα που ενεκρίθησαν χθε. Όχι. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Ο Πρόεδρος έλαβε από την ομάδα των Σοσιαλιστών ορισμένες αποφάσεις για να ανατροποποιηθούν κάποιες ε, θέσεις της αντιπροσωπείας. Οι αποφάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στα σημερινά πρακτικά και θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία ανακοίνωσή του. Και τώρα, το επόμενο θέμα στη μέρη διάταξη είναι επίκαιρη συζήτηση κατά πολέμηση του καρκίνου. Σας πληροφορώ ότι για τη συζήτηση αυτή δεν θα προβληθεί διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων, catch the eye και δεν θα γίνουν δεκτές μπλε κάρτες. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση και θα ήθελα να, δώσω το λόγο στον κύριο Βέμπερ που είναι ο συντάκτης. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπο του Συμβουλίου, πάνω από 40% των ε, συμπολιτών μας και το 40% και των παρόντων εδώ στην αίθουσα θα, κάποια στιγμή θα ασθενήσω από καρκίνο. Και αυτό σημαίνει απόγνωση. Ορισμένοι δεν θέλουν να το δεχθούν. Δεν ακούς τους γιατρούς, αρνείσαι την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά ξέρεις ότι ένα στους δύο καρκινοπαθείς ε, πεθάνουν, πεθαίνουν από το καρκίνο. Αισθάνεσαι χωρίς καμία δυνατότητα να αντιδράσεις. Αυτά είναι τα συναισθήματα που προκαλεί ο καρκίνος. Γι' αυτό το ερώτημα που θέτουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το εξή τρει, από τους τέσσερις Ευρωπαίους με βάση τις δημοσκοπήσεις ζήτησαν να γίνει βασική προτεραιότητα της Ευρώπης κατά πολέμηση του καρκίνου. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα των συμπολιτών μας. Οι Ευρωπαίοι ε, ε, ερευνητέ μας έχουν δείξει τι μπορούμε να επιτύχουμε. Για παράδειγμα, ο καρκίνος στους ε, ε, Έχει ποσοστά ίεσης 80% μαζί με διάφορους ε, επιφανείς ερευνητές από τα μήκη και τα ε, πλάτη της Ευρώπης υποβάλαμε ένα βασικό σχέδιο, ένα master plan για να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη, αγαπητοί συνάδελφοι, ο καρκίνος είναι περίπλοκη ασθένεια και έχει αμέτρητες μορφές εκδήλωσης. Για τα παιδιά, για παράδειγμα, κάθε χρόνο έχουμε 40.000 περιπτώσεις ιδιαίτερα σπανίων καρκίνων. Η Ευρώπη, αν συνεργαστούμε, λόγω των πολλών περιπτώσεων που έχουμε, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη επιτυχία εάν συνεργαστούμε. 18.000 ογκολόγοι, 15.000 ειδικά κέντρα ερεύνης και πολλά κέντρα έρευνας, 79 πανεπιστημιακές σχολές ασχολούνται με το θέμα αυτό. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Έτσι θα είμαστε πιο επιτυχημένοι. Η καθηγήτρια Αγγέλικα Έκαρτ από το Πανεπιστήμιο Σαριτέ του Βερολίνου μου έγραψε μια επιστολή που λέει ότι αν είμαστε φιλόδοξοι σε 10 χρόνια θα μπορούσαμε να θεραπεύουμε 9 από τα 10 παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Και ο καθηγητής Thierry Φιλίπ από το Παρίσι συμπλήρωσε ο συνδυασμό ε, έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και με προσωποποιημένη αντιμετώπιση μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό επιβίωση των ε, ασθενών 100%. Αυτά είναι εφικτά και πρέπει να τα επιτύχουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μια κοινή πολιτική πρόληψη του καρκίνου. Πρέπει να αποφεύγεται λοιπόν ο καρκίνος. Δεύτερον, όλα τα στοιχεία που έχουν ε, οι τράπεζες δεδομένων σε εθνικό επίπεδο να περάσουν σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων για τον καρκίνο. Επίση, θέλουμε μια στρατηγική για την έγκαιρη διάγνωση. Να επιτιθέμεθα στον καρκίνο εγκαίρω και να μην αφήνουμε κανέναν κατά μέρου. Ιδιαίτερα στι χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη, σήμερα οι καρκινοπαθεί έχουν 30% πιθανότητα να θεραπευθούν λιγότερο από ό,τι στι χώρε Δυτική Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση είναι απόλυτα απαράδεκτη σε μια Ευρώπη. Γι' αυτό με σύγχρονε μορφέ τηλεϊατρική θα έπρεπε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη να αυξήσουμε κατά πολύ τι πιθανότητε των ασθενών. Και να σκεφτούμε επίση και του συγγενεί των καρκινοπαθών. Πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία που να ασχολείται με τη φροντίδα των συγγενών. Το κόμμα μας θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει. Έχουμε μια νέα εντολή από του πολίτε τη Ευρώπη Τώρα εναπόκειται σε εμά να σημειώσουμε πρόοδου. Γι' αυτό, ω Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Θέλουμε όχι μόνο να γίνει σήμερα μια συζήτηση, όχι περισσότερο να θέσουμε προτεραιότητες σε αυτό το master plan, θα πρέπει με βάση τις μέχρι τώρα εργασίες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε στο μέλλον να υπάρξει μια ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου η οποία να ασχοληθεί με τη στρατηγική καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτό είναι το αίτημά μας και θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε και τώρα να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Η κυρία Τουπουράινεν, η ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Είναι τιμή που απευθύνομαι σε εσά για να συζητήσουμε την καταπολέμηση του καρκίνου στα πλαίσια αυτή τη επίκαιρη συζήτηση. Νομίζω είναι η κατάλληλη συγκυρία γι' αυτό. Τα πρόσφατα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο καρκίνος ε, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πρόκειται να γίνει ο πρώτος ε, λόγος θανάτου γιατί μειώνεται η θνησιμότητα από καρδιαγγειακές ασθένειες. Και από ό,τι φαίνεται η υψηλή θνησιμότητα δεν σχετίζεται με τους παράγοντες κινδύνου αλλά μπορεί να συσχετίζεται με την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όπως ξέρουμε, ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που συνήθως ε, χτυπάει ηλικιωμένους επειδή λοιπόν εμείς έχουμε υψηλότερο, ε, υψηλότερη μακριζωία, γι' αυτό ε, έχουμε περισσότερες περιπτώσεις ε, καρκίνου. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε μυρολάτρες ή πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αποφασιστικά. Η Προεδρία μας πιστεύει ότι οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και οι συμπολίτες μας να είναι στο κέντρο